24 δις ευρώ. Αυτός ε, είναι ο αριθμός ε, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ισχύει λοιπόν το εξής το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την Γραφειοκρατία στα 27 κράτη-μέλη. Το δίκαιο αυτό ε, του αναλογεί το 50% και η εθνική νομοθεσία καταλαμβάνει τα υπόλοιπα 50% ή 60%. Έτσι σε γενικές γραμμές αυτή είναι η συζήτηση για τα ποσοστά, αλλά σας ανέφερα και αυτή την τάξη μεγέθους για να έχετε έτσι μια εικόνα. Αυτό λοιπόν το ε, οικονομικής φύσεως θέμα γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Σήμερα ανοίγοντας ε, την εφημερίδα ε, και βλέποντας τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρεται στην αρτηριοσκληρωτική Ευρώπη που δεν παρουσιάζει πλέον καμία ανάπτυξη και κυριαρχεί κυρίως η γραφειοκρατία. Αν δούμε τι είπε εχθές ο Κάμερον στο συνέδριο του κόμματό του, θα ακούσατε ότι προανήγγειλε την ε, καταστροφή της Ευρώπης, ε, την ε, παρακμή της ε, Μεγάλης Βρετανίας και όλα αυτά οφείλονται στην γραφειοκρατία. Ακόμα και η καγκελάριος, η κυρία Μέρκελ και αυτή περίπου λέει τα ίδια. Άρα γενικότερα όλοι διαμαρτύρονται, αλλά οι άνθρωποι κάπου έχουν την αίσθηση ότι όλοι αυτοί οι ψηλόβαθμοι πολιτικοί καταγγέλουν την γραφειοκρατία, αλλά στη τελική ανάλυση δεν κάνουν τίποτα ίσως να γίνεται κάτι, αλλά οι πολίτες ε, δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Δεν γνωρίζουν ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και κάτι άλλο. Η γραφειοκρατία είναι σημαντική, διότι Υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της Ευρώπης και αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αισθάνονται ότι κατακλείζονται από αυτή την πλημμυρίδα των διατάξεων. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τους, ε, τις προσκαλέσαμε καταρχήν στη Λισαβόνα, εκεί όπου συνεδριάσαμε. Ε, προσκαλέσαμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις Αζόρες και από τη Γερμανία. Και να σας πω ένα παράδειγμα, στη συνεδρίασή μας της 3 η Μαου μία μικρή επιχείρηση από το ΑΑΧΕΝ η οποία κατασκευάζει πολύ ποιοτικά ε, μεγάφωνα μουσικής από πέτρα, μάρμαρο και γρανίτη αυτή η μικρή επιχείρηση δήλωσε ότι είναι απελπισμένη ε, διότι υπάρχουν όλες αυτές οι διατάξεις ε, περί προστασίας του περιβάλλοντος και πέρα από αυτές εκλήθη να καλύψει και άλλες διατάξεις που έχουν σχέση με το δίκαιο περί καταχώρησης, επισήμανσης και δηλώσεων. Επιπλέον υπάρχει και ένας άλλος νόμος που αφορά ε, τις ε, μπαταρίες, υπάρχει ο κανονισμός για τη συσκευασία, ο κανονισμός REACH, ο κανονισμός περί της επισήμανσης με το CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτές, ε, όλες αυτές οι διατάξεις που αφορούν και πέρα από αυτό ε, κάθε χρόνο να υποβάλλεται μια εγγύηση για τη χρηματοδότηση της απόσυρσης. Κάθε μήνα και κάθε χρόνο να δηλώνει κανείς τα προϊόντα που πούλησε ακόμα και αν είναι μηδενική η δήλωση. Αυτά όλα σας τα λέω έτσι ενδεικτικά. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Είπε, μάλλον εγκαταλείπω. Δεν κερδίζω τόσα πολλά χρήματα έτσι ώστε να μπορώ να καλύψω όλες αυτές τις ε, προδιαγραφές ε, μόνο με δύο-τρεις ανθρώπους. Και μόνο αν καταφύγω σε έναν ειδικό ε, φοροτεχνικό, ο οποίο ε, βεβαίω απαιτεί εκατοντάδε ευρώ, μόνο έτσι θα μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτέ τι ε, προποθέσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρησή του, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ο συγκεκριμένο άνθρωπο τώρα είναι αρκετά ευχαριστημένο γιατί μπόρεσε να τα καταφέρει. Βλέπετε όμω ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια άλλη παρατήρηση που αφορά στην πολιτική πτυχή της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Θα αφήσουμε καταρχήν κατά μέρος το θέμα της κρίσης που μαστίζει την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, η ε, πίεση σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων εξακολουθεί να είναι η βασική αιτία του γιατί η Ευρώπη δεν γίνεται αποδεκτή στα 27 κράτη-μέλη. Φαντάζομαι θα ρίχνετε καμιά ματιά στο ευρωβαρόμετρο και θα έχετε διαπιστώσει ότι φέτο την Άνοιξη το τελευταίο ευρωβαρόμετρο αναφέρει ότι όσον αφορά στο ερώτημα που έτσι στους πολίτες πώς αντιμετωπίζεις την Ευρώπη, οι απαντήσεις στη Γερμανία ήταν 43% Αυξήθηκε το ποσοστό, 43 λοιπόν ε, της απάντησαν σε αυτή την ερώτηση ότι η Ευρώπη είναι ε, ομολόχτης ε, γραφειοκρατίας και μας φέρνει μόνο επιβαρύνσεις. Το ίδιο περίπου ποσοστό είναι και στην Αυστρία, στις χώρες Μπενελούξ, στην Μεγάλη Βρετανία και στις σκανδιναβικές χώρες. Και σας είπα, τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από το 43% μέχρι το 50%. σε μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 50% των πολιτών που ε, έχουν σχέση με την Ευρώπη, απήντησαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η γραφειοκρατία και η επιβάρυνση για μας από τη γραφειοκρατία. Παρότι λοιπόν η Ευρώπη αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, η ουσία είναι ότι η πολιτική συζήτηση στα κράτη-μέλη, η πολιτική αυτή συζήτηση γίνεται μόνο ε, αφού έχουν ληφθεί καταρχήν οι βασικές αποφάσεις Βρυξέλλες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ε, και σε διεθνές επίπεδο ε, προσπαθούν να δουν τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Εδώ λαμβάνονται αποφάσεις και το μόνο που μπορεί να γίνει εκ των υστέρων είναι κάποιες διορθώσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί κανονισμοί οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί από τους ε, Θα σας αναφέρω και πάλι ενδεικτικά ένα παράδειγμα για τους ε, νέους οικονομικούς λαμπτήρες ή αν θέλετε για τις ε, προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει την κατανάλωση νερού με νέες μπαταρίες που θα τοποθετούνται στα μπάνια. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι τώρα στη Γερμανία που είναι η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γερμανία λοιπόν προσπάθησα να υπολογίσω πόσες ε, νομοθετικές ε, διατάξεις ε, ελήφθησαν τα τελευταία πέντε χρόνια, μετρήσαμε δηλαδή από το 1999 μέχρι το 2005. Πόσες λοιπόν νομοθετικές, νέες νομοθετικές διατάξεις επηρέασαν την οικονομία ή τους πολίτες. Αυτό δηλαδή σημαίνει όχι μόνο νόμους, αλλά και όπως σας είπα πράξεις και διατάξεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είχαμε πάνω από 21.000 νομοθετικές ρυθμίσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Και θελήσαμε να δούμε αυτές τις 21.000 πώς κατανέμονται σε Βρυξέλλες και Εθνικά Κοινοβούλια. Και με προς μεγάλη μας έκπληξη ε, οι 18.000, δηλαδή το 85% προέρχονται από τις Βρυξέλλες και μόνο οι υπολοιπόμενες 3.000 νομοθετικές ρυθμίσεις εκπονήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τις ε, εισηγήσει, πολύ λίγες υπήρχαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολλές εισηγήσει ε, για τα κρατημέλη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό πρόβλημα είναι. Ένα άλλο σημαντικό αίτιο για την αύξηση των ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων, κυρίως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας τροφίμων, ένα άλλο λοιπόν σημαντικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις στα 27 κράτη-μέλη και αυτές αντικαθίστανται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό βέβαια, πρέπει να το πούμε, διευκολύνει τις επιχειρήσεις, το ζητάνε αυτό οι επιχειρήσεις και έτσι προκύπτει και όλο μεγαλύτερη πίεση για προσαρμογή. Γιατί τελικά η Ευρώπη ε, θεσπίζει προσαρμογές που είναι απαραίτητε για την κοινή αγορά. Από την άλλη όμως δημιουργείται το πρόβλημα ότι οι πολίτες ενημερώνονται πολύ καθυστερημένα για το τι ακριβώς διαδραματίζεται στις Βρυξέλλες. Μόνο δηλαδή εφόσον το κράτος ή η περιφέρεια καλούνται να εφαρμόσουν αυτές τις ε, διατάξεις. Ενιαίες ε, ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις είναι βέβαια καθοριστικές για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά τα βλέπει κανείς στη συζήτηση που γίνεται για τις χημικές ουσίες, για τον κανονισμό REACH. Αυτό εμφανίζεται, έρχεται και επανέρχεται. Δηλαδή ο κανονισμός REACH ναι μεν καθορίζει διεθνή πρότυπα σχετικά με τις ε, χημικές ουσίες, πρότυπα που είναι σύγχρονα, που είναι προσαρμοσμένα στα αμερικανικά, ε, η Κίνα, ε, και αυτή λαμβάνει υπόψη στο τι θεσμοθετεί ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που έχει την έδρα του στο Ελσίνκι. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος που είναι ότι ε, προκύπτει μεγαλύτερη γραφειοκρατία και πάλι όπως σας είπα πλήττει αυτή κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι άλλο που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι η συμπεριφορά των πολιτών όπως επίσης ε, και των επιχειρήσεων. Και εδώ πάλι ε, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Από τη μία πλευρά όλοι διαμαρτύρονται για την υπερβολική γραφειοκρατία. Από την άλλη όμως θεσπίζονται νέοι κανονισμοί για τη βελτίωση της ζωής. Και μόνο αυτό Πολλοί απαιτούν αυτούς τους κανονισμούς στην προστασία του καταναλωτή, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην προστασία του περιβάλλοντο. Η καθοριστική εικόνα δεν είναι ο ενημερωμένος πολίτης, αλλά ο πολίτης που προσπαθεί να προστατευτεί μόνος του. Και βεβαίω ο πολίτης αυτός ε, επιθυμεί να διευκολύνεται η ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν εδώ υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έχουμε χιλιάδες βουλευτών και χιλιάδες ε, γραφειοκρατών στα 27 κρατη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι αυτοί ασχολούνται σίγουρα με το να βελτιώσουν ε, το επίπεδο ζωής των ανθρώπων. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος. Ξεκινάω από το ότι μια νομοθετική ρύθμιση επιθυμεί να αντιμετωπίσει προβλήματα οι στόχοι κατ' ουσίαν σωστοί είναι, κυρίως ε, μετά τις καταστροφές και τις κρίσεις ε, λαμβάνονται πάρα πολλές αποφάσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και κάτι το οποίο ε, μου έκανε εντύπωση τα τελευταία πέντε χρόνια είναι κάτι που γίνεται παρουσιάζεται σε πάρα πολλές συζητήσεις εκτός του Κοινοβουλίου είναι το εξής. Σε τελική ανάλυση η γραφειοκρατία αφορά την ένταση ανάμεσα στην ελευθερία των ανθρώπων και την ε, αφενός και την ασφάλεια που ε, προσφέρει το κράτος αφετέρου. Ναι, μεν όλοι ε, διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία, αλλά η ασφάλεια απαιτείται όλο και περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν ότι όσον αφορά αυτό το δίπολο θα πρέπει να βρεθεί καλύτερη ισορροπία, ε, λιγότερη κατακυδεμόνευση ε, σε επίπεδο καθημερινής ζωής, να μην ασχολούμεθα τόσο πολύ με την καμπύλη του αγκουριού και το αλάτι στα κουλούρια, αλλά να ασχολούμεθα με πραγματικά ουσιαστικά θέματα. Θα ήθελα ε, ως βουλευτής να σας το πω αυτό, να το υποστηρίξω, διότι διαπιστώνω, κυρίως εδώ, στις Επιτροπές του Κοινοβουλίου, σε επιτροπές ε, του Συμβουλίου. Ας αφήσουμε λιγάκι κατά μέρο την Επιτροπή. Οποτεδήποτε πρόκειται για νέες οδηγίες και νέους νόμους, πάντα αναζητείται ένας πολιτικός συμβασμός. Η μένη υπέρ αυτού, η άλλη υπέρ του άλλου και σε τελική ανάλυση η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. Ε, μερικές φορές λαμβάνονται ε, μέσα στη νύχτα αποφάσεις στο Συμβούλιο και ε, τελικά σφυριλατείται ένα συμβασμός και όλοι χαίρονται. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Ε, όταν πρόκειται για ε, την επίτευξη συμβασμού, κατ' ουσίαν τα προβλήματα είναι τεχνικής φύσεως. Τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του συμβασμού, ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες και για την γραφειοκρατία, αυτό μέχρι τώρα δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, ναι μεν όλοι διαμαρτύρονται γενικά για τη γραφειοκρατία, αλλά πολύ συγκεκριμένα όταν το θέμα που ε, τίθεται να ε, προκύψει μια συγκεκριμένη οδηγία, αυτό που ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Ας πούμε, ε, μια οδηγία περί των σωματιδίων, αιωρούμενων σωματιδίων γίνεται η κουβέντα, αλλά ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες στην πράξη, αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο, δεν παίζει ρόλο. Και αυτό ισχύει και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά βέβαια ισχύουν μέχρι σήμερα και το τονίζω αυτό. Μέχρι σήμερα. Τούτο λοιπόν αποτελεί πρόβλημα και εγώ ως, θέλω να το δείξω σε εσά ε, που είσαστε βουλευτές. Σας λέω και πάλι λοιπόν, αυτό είναι ένα αέναο καθήκον, είναι σαν να χρησιμοποιεί κανείς ένα τρυπάνι για να τρυπήσει ογκώδης, ε, για να τρυπήσει Η ομάδα υψηλού επίπεδου παρακολουθεί το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επίσης διαπιστώσαμε ότι από το 2012 και εφ' ε, μπορεί να υπάρξει μείωση της ε, γραφειοκρατίας μέχρι το κατά 25%. Υπήρξε ήδη μία μείωση ε, για 8-9 χρόνια είχαμε μία ομάδα υψηλού επίπεδου υπό την δική μου την Προεδρία και έτσι σε αυτό το χρονικό διάστημα καταθέσαμε περίπου 300 προτάσεις που οδήγησαν ε, στην ε, εξοικονόμηση 41 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέτεινε την ε, θητεία αυτής της Επιτροπής μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Η τελευταία έκθεση που καταθέσαμε οδήγησε τον πρόεδρο της Επιτροπής, με τον οποίο συζήτησα χτες για μισή ώρα, να επεκτείνει και πάλι την διάρκεια, ε, τη θητεία αυτής της Επιτροπής μέχρι το τέλος της δικής του της θητείας, δηλαδή ε, μέχρι το 2014, 31 Οκτωβρίου του 2014. Αυτά για την Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου. Σας λέω λοιπόν αυτό το πρόγραμμα δράσης και σύντομα θα υπάρξει από αυτού μία έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το πρόγραμμα δράσης σε γενικές γραμμές έχει υλοποιηθεί η Κομισιόν θα εξηγήσει τι ακριβώς κάναμε εμείς και ποιες προτάσεις μας υιοθετήθηκαν, την εξοικονόμηση των 30 δις ευρώ που προέκυψε, τα 10 δις ευρώ βρίσκονται σε φάση διαβουλεύσεων. Τελικά λοιπόν η Επιτροπή θα σας ενημερώσει, θα σας πει ότι το πρόγραμμα δράσης που προέβλεπε ότι το 25% του κόστους ε, γραφειοκρατίας που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ότι πράγματι αυτό μπορεί να μειωθεί, εμείς ε, αυτό το στόχο μας τον ε, εκπληρώσαμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και γι' αυτό σας λέω, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Το τελευταίο που θέλω να σας πω αφορά στην παράταση. Για μένα ήταν απόλυτα σαφές, επειδή για πολλά χρόνια ήμουν υπουργό ετρικών, ε, πρωθυπουργό στη Βαβαρία, ε, είχα πάρα πολλές ε, κυβερνητικές θέσεις. Να σας πω λοιπόν το εξής. το ευρωπαϊκό επίπεδο δέχεται χτυπήματα χωρίς να μπορεί να αμυνθεί. Οι πρωτεύουσε της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν συνεχώς στις Βρυξέλλες οποτεδήποτε προκύπτει πρόβλημα γραφειοκρατίας. Και εγώ το έκανα αυτό. Όλοι λένε αυτοί οι χαζοί στις Βρυξέλλες ε, έχουν κάνει αυτό το λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, να απευθυνθείτε στις Βρυξέλλες και όχι σε εμά. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Γι' αυτό λοιπόν το 2011 κάναμε μία έρευνα για το πώς ακριβώς Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στα 27 κράτη-μέλη. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι περίπου το 1 τρίτο του γραφειοκρατικού άχθους που προκύπτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 1 τρίτο αυτό δεν προκαλείται από την Ευρώπη αλλά από την ε, ανελειπή, μάλλον από την ε, μη αποτελεσματική εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Κυρίες όμως, ε, σας λέω, από την μη αποτελεσματική εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις, να δούμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες. Είδαμε λιγάκι την διαδικασία ε, και τις ε, νομοθεσίες που αφορούν στους δημόσιους διαγωνισμούς και τις ε, κρατικές προμήθειες. 77 ημέρες ε, διαρκούν αυτές οι διαδικές στην ε, Λιθουανία, αλλά 44 μόνο στη Μάλτα. Συγγνώμη, 241 στη Μάλτα. Όσον αφορά το κόστος, 22 ε, εργάσιμες μέρες στο Λουξεμβούργο, ενώ 93 εργάσιμες μέρες στη Βουλγαρία. Άρα δηλαδή το μήνυμα που προκύπτει από αυτούς τους αθμούς είναι ότι σαφώς και μπορεί να υπάρξει βελτίωση. εγώ απευθύνθηκα στους 27 ε, πρωθυπουργούς των κρατών μελών και τους είπα για πέστε μου ένα παράδειγμα όπου είχατε πολύ καλή εφαρμογή ε, κοινοτικών διατάξεων και μου ανέφεραν ε, όλοι τις βέλτιστες πρακτικές. Αλλά οι βέλτιστες πρακτικές ε, συνεπάγονται και κακές πρακτικές. Εμείς λοιπόν κάναμε μία έρευνα, ε, φαντάζομαι ε, θα γνωρίζετε αυτό το εγχειρίδιο που φέρει τον τίτλο «Τι μπορεί να βελτιώσει η Ευρώπη». Συγκρίναμε λοιπόν 27 περιπτώσεις και βασικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να ξεκαθαρίσουν δηλαδή γιατί οι Γερμανοί τα πάνε χειρότερα από τους Γάλλους. Γιατί στην Αγγλία οι διαγωνισμοί αυτοί ε, είναι πιο χρονοβόροι από ό,τι στη Δανία. Και οι διαφορές είναι εντυπωσιακές. Σας λέω για άλλη μια φορά ότι θα μπορούσε κανείς να εξοικονομήσει 40 δι ευρώ που αφορούν στο γραφειοκρατικό άχθος και την επιβάρυνση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εάν ακολουθεί το παντού η ίδια βέλτιστη πρακτική. Ε, θα φέρω άλλο ένα παράδειγμα προς μίμηση. Στην Εσθονία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει νόμος που απαγορεύει να ξανασυγκεντρωθούν δεδομένα τα οποία ήδη έχουν συγκεντρωθεί ηλεκτρονικά και έχουν καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρό. Τι σημαίνει αυτό, ότι από τη στιγμή που άπαξ συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία, τέλος, μετά να πάνε όλοι να τα βρουν. Ε, αλλά στη Γερμανία ή στη Γαλλία συνέχεια ρωτάνε τους ανθρώπους, ζητάνε από αυτούς ε, στοιχεία, είτε το Υπουργείο είτε η υπηρεσία για τα καρτέλ, μα μία φορά να ζητάει το κράτος τα στοιχεία και μετά να τα οργανώνει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτός που θέλει στοιχεία να μπορεί να ψάξει να τα βρει σε ένα και μόνο φορέα. Πάμε στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία οι δημόσιοι διαγωνισμοί υποχρεωτικά γίνονται ηλεκτρονικά και η ψηφιακή συμμετοχή στην Πορτογαλία ξεπερνάει το 75% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι μόνο 5%. Πάμε στη Γερμανία. Υπάρχει ένα monitor που λέγεται ένας φορέας στη Γερμανία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στη Γερμανία έχουν πάρα πολλές φορές δυσκολίες να ενημερώνονται σωστά για τις ευρωπαϊκές ε, διατάξεις. Όμως τώρα στη Γερμανία υπάρχει το εξή σύστημα. Ο μικρομεσαίος έχει το φωτεινό σηματοδότη. Εκεί βλέπει τι προετοιμάζει η Ευρώπη. Όταν είναι κόκκινος λέει πρόσεξε σε αφορά. Το κίτρινο έτσι και έτσι και το πράσινο κανένα πρόβλημα. Άρα δηλαδή πολύ γρήγορα μπορεί κανείς να ενημερωθεί τι υπάρχει και τι ε, θα προκύψει από τις Βρυξέλλες για τον επιχειρηματία. Σας ε, ανέφερα λοιπόν το αποτέλεσμα. Και επιτρέψτε μου και μία άλλη παρατήρηση. Εχθές, το λέω ξεκάθαρα, πίστευα ότι ε, κάπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια γενική εποπτεία εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών. Ήμουν αφελή, το ομολογώ, ειλικρινά πολύ αφελης το ομολογω ειλικρινα πολυ αφελη και ρώτησα τον Υπουργό Εσωτερικών τη Γερμανία. Για πε μου, του λέω, αν κατασκευάζεται αυτός ο περίφημος ε, σιδηροδρομικός σταθμός της Ουτγάρντης, ο σταθμός 21 που έχει προκαλέσει πολλές φασαρίες, αν κατασκευάζεται στη Ρώμη, στο Εντιμβούργο, στη Γαλλία, οπουδήποτε, μου είπε, κοίτα Έντμουντ, <clears throat> Κανένα πρόβλημα, θα σου δώσω σε τέσσερις εβδομάδες τα στοιχεία γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει μελέτη. Έχουν περάσει 8 εβδομάδε, τίποτα δεν ξέρουμε. Ούτε καν τα δικά μα τα στοιχεία. Και σκέφτηκα, μα θα πρέπει να έχει τα στοιχεία τουλάχιστον η Κομισιόν. Έτσι, έστω κατά προσέγγιση μια σύγκριση. Ούτε και αυτή, τίποτα. Τίποτα, απολύτω τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα ε, το οποίο ετέθη ε, στην τελευταία στην διάσκεψη κορυφής ε, τον Ιούνιο και στο Συμβούλιο παρότι παράλληλα γινόταν η συζήτηση για το ευρώ οι αρχοί κρατών και κυβερνήσεων βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν με τη γραφειοκρατία και κατέληξαν στο ότι τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου οφείλουν να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες. Δηλαδή αν η Γαλλία έχει ήδη εφαρμόσει μία οδηγία ή η Αυστρία ακόμα δεν το έχει πράξει, τότε έχει νόημα ο αρμόδιος υπάλληλος της Αυστρίας να απευθυνθεί στους Γάλλους και να τους πει σας παρακαλώ πέστε μου πώς το κάνατε ακριβώς ε, ίσως ε, κι εγώ μπορώ να μάθω κάτι και να υιοθετήσω κάτι αυτή η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στις διοικήσεις των κρατών μελών αυτή η ανταλλαγή απόψεων σήμερα δεν γίνεται σχεδόν καθόλου και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μέλημα, ένα αίτημα που πρέπει να ε, εφαρμοστεί στο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα Impel, και εκεί υπάρχει ένα σχετικό εργαλείο, καλό αυτό το εργαλείο, υποκλίνομαι, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων επ' αυτού. Νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αν το Κοινοβούλιο ασχολείται με αυτό το σύστημα το δίκτυο Impel, όπως αναφέρεται. Καταλήγοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πάλι υποκλίνομαι, παρακολουθώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διοίκησή της εδώ και περίπου 30 χρόνια. Και τότε ήμουνα ε, νέος υφυπουργό και συζήτησα με τον Ζακ Ντελόρ για τα θέματα της ε, επικουρικότητας. Αυτό το θέμα είναι πανάρχαιο, αν θέλετε. Πάντως διαπιστώνω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε χώρα αλλαγή νοοτροπίας. Σήμερα δηλαδή, κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου οδηγίας, σκέφτονται πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 10 χρόνια τις επιπτώσεις. Υπάρχει το περίφημο περίφημο Impact Assessment Board, αυτό το όργανο το οποίο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Καμία αμφιβολία από αυτού, αλλά νομίζω ότι οι γενικές διευθύνσεις ήδη σκέπτονται ποιες θα είναι επιπτώσεις. Και διαπιστώνω ότι στην Επιτροπή πολλοί σκέπτονται ότι ναι μεν έχουμε τώρα ένα συμβασμό, όμως αυτός ο συμβασμός θα πρέπει να πάει στο Κοινοβούλιο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Ίσως τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο περίπλοκα, θα πρέπει να αναζητηθεί νέος συμβιβασμό και μέχρι τώρα το ε, Κοινοβούλιο εντάξει, δεν πολύ σκέφτεται το θέμα των ε, γραφειοκρατικών συνεπειών. Τώρα όμως διαπιστώνω ότι και στο Κοινοβούλιο έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας ενημέρωσε στην ε, ομάδα μας σχετικά με τη σύσταση μιας γενικής διεύθυνσης που θα ασχολείται με μελέτες αντικτύπου. Αυτή η Γενική Διεύθυνση θα επανδρωθεί με 30 συνεργάτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχολείται και αυτό με τις ε, συνέπειες ε, που θα προκύπτουν από μια οδηγία. Και δεν θα περιορίζονται μόνο σε αυτά που λέει το Impact Assessment Board της Κομισιόν. Ε, θα ασχολείται και το Κοινοβούλιο. Αυτό λοιπόν το βρίσκω ιδιαίτερα θετικό και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γνωρίζω και την έκθεση Νίμπλερ, τη σχετική. Όποιος, ε, μάλλον αυτός που είναι λιγάκι επιφυλακτικός, ε, είναι το Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο σκέπτεται να συστήσει και αυτό. Μια ομάδα που θα ασχολείται με μελέτες αντικτύπου που θα υπάγεται στον ίδιο τον κύριο Φαν Ρομπέι. Άρα δηλαδή σύντομα θα έχουμε τρεις φορείς, Κομισιόν, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο που θα ασχολούνται με μελέτες αντικτύπου. Ε, μπορεί κάποιος να φανταστεί και γιατί να έχουμε τρεις και να μην έχουμε μόνο μία. Δύσκολο αυτό. Ίσως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο οι τρεις θεσμοί, όπως σας είπα, να ασχολούνται με μελέτες αντικτύπου, με την ε, αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, γιατί μέσα από τον ανταγωνισμό αυτόν κάτι καλό θα προκύψει. Τελευταία παρατήρηση κυρίε και κύριοι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ε, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Αγωνίστηκα να παραταθεί η διάρκεια ζωής της Επιτροπής μου και τώρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου Υπάρχουν ε, δύο θέματα που μας απασχολούν αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις πολύ μικρές μάλιστα, οι οποίες λόγω της γραφειοκρατίας επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από τις μεγάλες που έχουν τη σχετική υποδομή για αντιμετώπιση της. Οι μικρομεσαίες είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης. Ε, με βάση εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εφέτος ε, θα ε, τύχουμε δυστυχώς ε, μηδενική ανάπτυξη, ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη θα ανέρχεται στο 4%. Η Ευρώπη σιγά σιγά, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ε, προβάλλεται η επιχειρηματικότητα και να μην αναχαιτίζεται αυτή από υπερβολική γραφειοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν ε, η ομάδα υψηλού θα επιληφθεί του θέματος. Η γραφειοκρατία που επιβαρύνει κυρίως τις ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι πρόβλημα. Και βεβαίως και οι διοικήσει των κρατών μελών καλούνται να εργάζονται αποδοτικότερα, διότι η διαφορά στην αποδοτικότητα των διοικήσεων των κρατών μελών. Θα είμαι εδώ λιγάκι προσεκτικός. Θα πω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή και μερικά κράτη έχουν τεράστια προβλήματα να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης. Η Κομισιόν λοιπόν τα επόμενα δύο χρόνια θα σκεφτεί το θέμα αυτό και έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται τώρα σε μια επικοδομητική διαμάχη με τις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών. Εχθές ε, ο πρόεδρος, όπως σας είπα, σκέφτηκε να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας φορέας τεκμηρίωσης, ο οποίος θα ασχολείται με την εφαρμογή την υλοποίηση των κοινοτικών ε, οδηγιών. Αυτό είναι μια νέα τάση που φαντάζομαι σας ε, εξυπηρετεί, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς πολύ συχνά δέχεστε διαμαρτυρίες για τις οποίες δεν φέρετε εσείς την κύρια και κέρια ευθύνη. Ε, η ευθύνη οι αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν κατά την εφαρμογή. Αυτοί όμως που πλήττονται παραπέμπουν μάλλον οι αρμόδιοι παραπέμπουν στις Βρυξέλλες για να απεκδίονται των ευθυνών τους και θεωρώ ότι είναι αστείο το γεγονός ότι ο πρώην ε, Πρωθυπουργό ε, της Βαβαρίας ως ε, υπέρμαχος της Ομοσπονδιακής Διακυβέρνησης σε τελική ανάλυση τώρα κατηγορεί τους πρώην συναδέλφους του ότι αυτοί φταίνε, ότι αυτοί είναι πολύ αργοί στην εργασία τους. Αυτό όμως είναι ένα θέμα δικό σας που απασχολεί κυρίως εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εγώ προσπάθησα να σκιαγραφίσω λιγάκι την κατάσταση και όποιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ίσως μπορεί να διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει την εφαρμογή, την εκτέλεση των διατάξεων. Την επόμενη και μεθεπόμενη εβδομάδα ε, θα παρίσταμε στην διευρυμένη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πολλοί συνάδελφοί μου από την ομάδα υψηλού θα πάνε αντίστοιχα στο Σουηδικό, Ιταλικό, Δανέζικο Κοινοβούλιο και θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση, έστω να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για το τι μπορεί κανεί να κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα περιζόταν και οι, τα εχθρικά συναισθήματα απέναντι στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς ε, για την πολύ ζωντανή ε, παρουσίασή σας γιατί ε, έριξα έτσι μια ματιά στην αίθουσα και όλοι κρέμονταν από τα χείλη σας. Είπατε βέβαια και πολλά και προκλητικά και αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο διότι αναφέρατε στην ομιλία σας ορισμένα θέματα τα οποία σίγουρα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον. Εσείς μιλήσατε για την εφαρμογή των διατάξεων. Εγώ είμαι εισηγητής για το backloading, ε, την καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστημα ε, εμπορίας, ποσοστώσεων εμπορίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Γερμανία πρέπει να καταβάλει 35 ευρώ ε, για αυτό το πιστοποιητικό, ενώ στη Γαλλία μόνο 26. Ε, κοινή αγορά είναι. Αλλά και έχουμε και την επέτειο, αλλά βλέπετε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφορές. Δεν υπάρχει μια γενική επισκόπηση του πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις. Και εγώ ε, θορκιζόμουνα ότι τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει πώς ακριβώς εφαρμόζονται οι διατάξεις. Οποτεδήποτε έρχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μιλήσει για την εφαρμογή ε, ευρωπαϊκού δικαίου, εδώ προκύπτουν πολλές ε, και έντονες συζητήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Ο κύριος Ζήμπα έχει ζητήσει το λόγο. Είναι ο συντονιστής, ένας από τους ε, συντονιστές του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίως ευχαριστούμε για την ε, πρωτοβουλία που, ανέλαβε, που αναλάβατε να καλέσετε εδώ τον κύριο Στόιμπερτ. Ε, κύριε Στόιμπερ, πρέπει να πω ότι με μεγάλη μου χαρά σας άκουγα και παλαιότερα όταν ήσασταν ε, Πρωθυπουργό. Ακούγοντας αυτά που μας είπατε σήμερα ε, πρέπει να πω ότι τελικά αλλάξατε πλήρως γνώμη γιατί όταν ήσασταν Πρωθυπουργό της Βαβαρίας τότε κι εσείς υψώνατε το δάκτυλο κατά της, των Βρυξελών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τέλος πάντων, τα πράγματα άλλαξαν, αλλάξατε τελείως. Επειδή και βέβαια είσαστε βαβαρός, ε, φαντάζομαι ότι δεν θα με παρεξηγήσετε που θα είμαι ειλικρινής. Ω βαβαρό έχετε συνηθίσει σε ειλικρινεί κουβέντες. Κύριε Στόιμπερ, αυτό που δεν είπατε όμως είναι ότι οποτεδήποτε θεσπίζεται ευρωπαϊκή διάταξη, κατ' ουσίαν η διάταξη αυτή αφορά 27 κράτη-μέλη και δεν ε, θεσπίζουμε 27 μεμονωμένες διατάξεις. Εσείς λοιπόν έρχεστε, έρχεστε από ομόσπονδο κράτος και εγώ έρχομαι από ομόσπονδο ε, κράτος. Στην Αυστρία ας πούμε έχουμε 9 διαφορετικές διατάξεις για τα σανσέρ. Άλλες οι διατάξεις για τη Βιέννη, άλλοι ε, οι ρυθμίσεις ασφαλείας για τη Βιέννη, άλλες για το Τυρόλο ξέρω εγώ. Άρα δηλαδή πρέπει να πλασιάσετε, 27 συν ε, πόσα είναι τα μόσποντα, οι ομόσπονδες ρυθμίσεις και η Βαβαρία και για τη Βαβαρία ισχύει αυτό άρα σας παρακαλώ να το έχετε αυτό κατά νου γιατί ε, οι υπολογισμοί που κάνατε Καλά ακούστηκαν, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας πει τι σημαίνουν αυτά. Να σας πω εγώ τι σημαίνουν, θα σας τα πω ξεκάθαρα. Τίποτα, καινή αριθμή. Γιατί εκείνο που πρέπει να υπολογίσετε είναι ότι αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, πόσο θα κόστιζε αυτό. Και εκεί τα ποσά θα ήταν ανυπολόγιστα, τεράστια. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που είπατε και τώρα Better Europe, καλά τα λέτε, εντάξει συμπαθητικά, αλλά τίποτα δεν είναι και αυτό τίποτα δεν είναι. Το ότι πρέπει να βελτιωθούν ορισμένα πράγματα, αυτό είναι αναμφίβολο. Έρχεται τώρα και ένα άλλο πρόβλημα ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση που το ε, καλλιεργούν πάρα πολλοί συνάδελφοι μόνο που σε τελική ανάλυση όλοι μετακυλίουν την Ευρώπη πάνω την δεύτερη Ευρώπη και μπορώ ε, να σας αναφέρω χιλιάδες παραδείγματα όπου η Ευρώπη δέχεται τις επιπλήξεις χωρίς να φταίει. Εσείς ας πούμε μιλήσετε για λαμπτήρες. Κοιτάξτε υπήρξαν πάρα πολλές αποφάσεις. Υπουργοί περιβάλλοντος. Ακόμα και ο Γερμανός ε, υπουργό ε, και στη Γερμανία και στην Αυστρία έγινε τεράστια συζήτηση μόνο που σας παρακαλώ πάρα πολύ πέστε μου έναν πολιτικό από τη Γερμανία και έναν από την Αυστρία που να είχαν το κουράγιο να υπερασπιστούν την άποψή τους. Ε, δεν ξέρω πώς τους λέτε λύση οπωσδήποτε αλλά εμείς ήμασταν εκείνοι που εισαγάγαμε αυτούς τους κακούς λαμπτήρες. Το ότι όμως έχει νόημα ε, να στηρίξει κανείς αυτούς τους λαμπτήρες, να δημιουργήσει θέσεις ε, πράσινης απασχόλησης. Ε, αυτό η Γερμανία πού ήτανε, πού ήταν η Γερμανία, πουθενά. Το λέω λοιπόν ξεκάθαρα. Άρα δηλαδή βασικό πρόβλημα είναι το θέμα της επικοινωνίας. Και μόνο αυτό, αλλά το λέω και ξεκάθαρα, η δηλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών και των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Να πούνε ότι κοιτάξτε οι ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται σωστά. Και τώρα με συγχωρείτε κύριε Στέμπρα, αλλά είμαι αναγκασμένο να μη διάσω. Εσεί έρχεστε από κράτο μέλο και εγώ έρχομαι από άλλο κράτο μέλο ε, που έστειλαν επιστολέ ε, στι Βρυξέλλε. Τώρα ε, θέλουμε να φτιάξουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θέλουμε να περιορίσουμε το κόστο. Έχουμε 6% διοικητικό κόστο και η πολιτική στη Γερμανία και αυτή στην Αυστρία από όλε τις, ε, τα πολιτικά κόμματα λένε ότι πρέπει να εξοικονομηθεί το κόστο από το προσωπικό. Και όλοι αυτοί που οι διερμηνεί που βρίσκονται εδώ που είναι αναγκασμένοι να μιλάνε τα κακά τα δικά μου τα αυστριακά από αυτού να του κόψετε 2 ε, ή 3%. Εντάξει, κόψτε του διερμηνεί και α μιλάμε όλοι αγγλικά. Ε, δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε. Η Ευρώπη είναι ένα περίπλοκο πράγμα και κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Ε, αν θέλετε να έχουμε μόνο μία γλώσσα, ε, να μην έχουμε 22 διαφορετικέ γλώσσε και για να δούμε αν αυτό θα γίνει αποδεκτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η δέσμευση, κανεί δεν αναλαμβάνει τι ε, πολιτικέ ευθύνε για αυτή την Ευρώπη. Περί αυτού πρόκειται και πρόκειται επίσης και για θέματα επικοινωνίας. Διότι και τώρα απευθύνομαι σε εσά σε συγκεκριμένα κύριε Στόιμπερ. Εντάξει, καλό αυτό που κάνετε, αλλά κάπως πρέπει και να το ανακοινώσετε, να το διαδώσετε. Ε, το λέτε σε εμά, σε εμάς εδώ, ε, έτσι κι αλλιώς εμείς ε, πεπισμένοι είμαστε. Να πάτε στη Βαβαρία, στη Πυραρία, εκεί να πάτε, στο σπίτι σας. Τώρα είχατε Οκτώμπερ και αυτά που είπατε εδώ να πάτε να τα πείτε στη Βαβαρία. Για πηγαίνετε, για να δούμε. Όχι, για πηγαίνετε. Και σας παρακαλώ ε, μπροστά στον Πρωθυπουργό σας, τον κύριο Ζέχοφερ, και για να δούμε τι θα γίνει, να το πείτε μπροστά στους συναδέλφους σας στη Τσέσου. Γιατί αν έχετε το θάρρος, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα σας χειροκροτήσει. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα εδώ μια χαρά, πολύ ωραία, συζήτηση σε διανοούμενους, μόνο επί της ουσίας. Κοιτάξτε, η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση γίνεται στα 27 κράτη-μέλη και εκεί κανείς δεν έχει το θάρρος να αντικρούσει την κοινή γνώμη. Ε, το βλέπετε αυτό στον προπολογισμό. Να γίνουν περικοπέ και λέτε η Κομισιόν, να τα κάνετε και η Κομισιόν. Ε, με τι να κάνει η Κομισιόν. Και εμεί συνεχώ την επικρίνουμε την Κομισιόν και καλά κάνουμε. Μόνο που πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι τη Κομισιόν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, έχουν κίνητρα και έρχεται εσεί εδώ και λέτε αυτοί δεν έχουν πίνακε. Ε, με συγχωρείτε. Άμα ζητάμε τους, όταν ζητάμε του πίνακε από την Κομισιόν, ξέρετε τι λένε και τα κρατημένα του Συμβουλίου. Αποκλείεται. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το Συμβούλιο δεν θέλει να έχει ε, Ευρώπη, αλλά όλο βρίζει που τα κράτη δεν προσαρμόζονται σε ευρωπαϊκά μοντέλα. Ε, να έχετε το θάρρος λοιπόν και κυρίως εσείς ως πρώην Πρωθυπουργό Κρατηδίου να το πείτε αυτό στους συναδέλφους σας, τον τώρα Πρωθυπουργό σας, να το πείτε στους Αυστριακούς πολιτικούς, στην Γερμανίδα Καγκελάριο, εκεί να πάτε να τα πείτε τελικά όταν θα έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, τότε εντάξει να δούμε λιγάκι τις λεπτομέρειες. Και κάτι άλλο πρέπει επίσης να πούμε, το κόστος της μη δράσης, non-action, αυτό που δεν οδηγεί. Τώρα, ε, όταν μιλάει κανείς ε, για την οδηγία περί καθαρότητας ε, της ατμόσφαιρας, κοστίζει και αυτό. Αλλά είδατε και πόσοι πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχει καθαρή ατμόσφαιρα. Και αυτό πανηρό δεν είναι. πρέπει να προσέξουν. Λυπάμαι πολύ που ήμουν έτσι συναισθηματικά φορτισμένος και παρασύρθηκα, αλλά τι να πω κι εγώ, αυτό το μήνυμα να πηγαίνει κανείς και να λέει τι λάθος κάνουμε εδώ και μετά στην πατρίδα του να διαφορετικά, ας πάρουμε το νερό. Λέτε ας πούμε πούμε ανεπαρκής ε, διοίκηση. Ας πούμε στην οδηγία περί διαχείριση Στο Τυρόλο όταν κατασκευάζεται μία μικρή μονάδα η, ο Εθνικός Φορέας λέει για να χρησιμοποιήσετε το νερό από το ριάκι, να πάτε να αφαιρέσετε τις πέτρες με το χέρι, χειρανακτικά. Αυτή είναι μία διάταξη, αυτή είναι μία πραγματικότητα. Δεν είναι θεωρητικό. Άρα δηλαδή αποτελεσματική διοίκηση τι σημαίνει αυτό. Στην ε, ε, Ελλάδα πολύ καλύτερη είναι η διοίκηση που λέει θέλετε νερό από το ριάκι, τι, ποιο χέρι και χρησιμοποιείτε χέρι, βάλτε εκεί το τρακτέρ και αποσύρετε τα όλα. Αυτή μπορεί να είναι καλύτερη διοίκηση. Υπάρχουν όμως, σας λέω, ότι ε, υπάρχουν και διαφορετικές παραδόσεις. Αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλετε εσείς δεν υπάρχουν. Σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ε, την άποψη ενός τυρολέζου και στο σπίτι μας να κοιτάμε τα του οίκου μας και όταν θα έχουμε δει τα του οίκου μας θα τα καταφέρουμε καλύτερα και εδώ. Πρόεδρος, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση που αφορά σε αυτά που είπε ο κύριος Ζέμπερ Κοιτάξτε, μην αντιμετωπίζετε εδώ ως κάποιον ο οποίος ε, είναι πρόεδρος ε, μιας επιτροπής επίτιμων μελών, επίτιμων μελών από διάφορα κρατημέλη, ε, ο οποίος θα πρέπει να λύσει τα πάντα. Και δεν άλλαξα τα ρούχα μου ως μανολιός και έγινα αλλιώ, όπως λέμε χαρακτηριστικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Υπήρξαν δύο πολιτικοί τη δεκαετία του 90 οι οποίοι ήταν κατά της ταχείας εισαγωγής του ευρώ. Εγώ ήμουν ο ένα και ο άλλος ο Γερμανός ο κύριος Μπίντενκοπφ. Γι' αυτό τώρα στη Γερμανία όλοι με αντιμετωπίζουν ως Θεό. Ε, επειδή ήμουνα κατά της ε, εισαγωγής ε, του ευρώ και σήμερα όμως είμαι υπέρ αυτού. Και ξέρετε γιατί. Δεν είναι επειδή σας είπα άλλαξα τα ρούχα μου και έγινα αλλιώ, αλλά διότι οι καταστάσεις άλλαξαν, άλλαξαν, άλλαξε το γίγνεσθε. Και όσον αφορά την επικουρικότητα, εγώ σας βοηθάω απλά. Εσείς καλείστε να κάνετε τη συζήτηση στα κόμματα και σε εθνικό επίπεδο. Σας είπα, αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο δέχεται ραπίσματα για πράγματα που δεν είναι αρμόδιο. Τα τελευταία χρόνια εγώ πάω σε όλες, σε πολλές εν πάση περιπτώσει, οικονομικές ενώσεις και λέω να, τα έχω κουβεντιάσει αυτά με τους αρμόδιους. Επίσης τα κόμματα, τα συζητάω, αυτά που μου είπατε εγώ τα κάνω, στο βαθμό του δυνατού βέβαια. Προσπαθώ να εξηγήσω ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Βρυξελών και πού μπορεί κανείς ε, να μιλήσει για αρμοδιότητες, ε, κατά πόσον ενδεχομένως θα πρέπει να δει κανείς διαφορετικά το θέμα. Κύριε Ζήμπα, ε, θα πρέπει ένα πράγμα να δεχτείτε σε αυτή την ευρωπαϊκή διαδικασία. Τη δεκαετία του 80, το αργότερο από το 86, έχουμε την ευρωπαϊκή πράξη ή τις ευρωπαϊκές πράξεις όπου και για τη διαχείριση υδάτων υπήρξε ε, χώριση αρμοδιοτήτων από τις Βρυξέλλες στα κράτη-μέλη και τη δεκαετία του 90 Υπάρχουν όλο και περισσότερα σημαντικά πράγματα ε, στο εταιρικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο, στο δίκαιο περί φαρμάκων, παντού. Οι άνθρωποι βέβαια αυτό δεν το συνειδητοποιούν, αλλά όλο και περισσότερο εκχωρούνται αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σήμερα αν εξαντλήσει τις αρμοδιότητες της ή εξαντλεί τις αρμοδιότητες της. Και εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να συζητάμε μόνο λεπτομέρειες, αλλά να συζητάμε και για το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει παντού επικουρικότητα. Σε γενικές λοιπόν γραμμές σας λέω το θέμα της ε, εφαρμογής της ε, εκτέλεσης του ε, κοινοτικού δικαίου Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εφόσον με προκαλέσατε κιόλας, να σας πω κι εγώ ότι υπάρχει η Ευρώπη των ελίτ, των, της αφρόκρεμας. Δεν γίνεται διαφορετικά και αυτές οι ελίτ δεν συμπαρέσυραν τους πολίτες. Απλά το διαπιστώνω αυτό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν κατ' ουσίαν. Ίσως αυτό να οφείλεται και σε εσά. Ε, ίσως, δεν ξέρω, δεν ξέρω, το λέω σου γενικά. Ίσως διότι οι ευρωβουλευτές δεν ενημερώνουν τόσο καλά τους πολίτες το τι κάνει η Ευρώπη. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά όσον αφορά τα θέματα, εγώ σας δίνω τα κίνητρα και εσείς είστε πολιτικός. Εγώ είμαι συνταξιούχος πολιτικός. Συγγνώμη. στο σύντομο χρονικό διάστημα που είμαι πρόεδρος αυτή ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ο κύριος Ζιμπ ε, ξελέγει πριν από λίγο ο καλύτερος βουλευτής ε, της ε, ομάδας περιβάλλοντος. Ο κύριος Γιολάν έχει το λόγο. Äh, Χαίρομαι που σα έχουμε μαζί σα σχεδόν ποτέ δεν έχω δει το Ζέμπερ να χάνει την ε, ηρεμία του και την ψυχραιμία του όπως σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ο... νομίζω ότι έσπασε όμως ένας πάγος, έτσι, και τώρα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ακούστε, εδώ είμαστε περισσότερο από 700 ευρωβουλευτές, υπάρχουν 70.000 εθνικοί βουλευτές αν λένε ανοησίες 70.000, πώς θέλετε να διορθώσουμε την κατάσταση εμεί οι 700. Τέλος πάντων, είμαστε σε μία περίοδο συνεχών αλλαγών. Και βεβαίω, εάν δούμε το όλο θέμα σφαιρικά, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Εσείς, καθώς και άλλοι συναδελφοί σας, εθνικό επίπεδο, λέτε ότι όταν εγκρίνεται μία νομοθετική πράξη στο Βερολίνο είναι πολιτική και όταν γίνεται στις Βρυξέλλες ότι είναι γραφειοκρατική ε, και διοικητική απόφαση. Αυτό είναι το λάθος κατά την άποψή μου. Δεδομένου ότι εμείς εγκρίνουμε εδώ νομοθεσιτικές πράξεις για να γίνει πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική, καλύτερη η Ευρώπη, για να μπορέσουν να γίνουν νέες βιομηχανίες πιο ανταγωνιστικές. Φανταστείτε, αν δεν είχαμε τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σλοβενία, η Γερμανία και άλλες χώρες, θα έπρεπε η καθεμία να εργάζεται και αναπτύσσεται μόνη της και θα είχαμε μεγάλη οπισθοδρόμηση. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι λίγο γελία. Και αυτά δεν έχουν σχέση με την ε, δημοκρατία. Ας αναφερθούμε στα οικονομικά θέματα. Ας πούμε κάτι άλλο. Ότι το τηλέφωνο του ντους δεν είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται και ενοποιείται σύμφωνα με την κοινωτική νομοθεσία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή να κάνουμε, να αρμονίσουμε τα πάντα για να γελιοποιήσουμε την Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρατε κάτι άλλο, το οποίο και εμείς πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Η μεταφορά στο κάθε εθνικό δίκαιο. Δεν υπάρχει μόνο η νομοθετική δουλειά μας, η οποία είναι σημαντική. Μιλήσατε, όπως είπε και ο Ματίας Γκρόσε, για το κόστος που είναι διαφορετικό για κάποια θέματα στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αλλά εάν δεν υπάρχει κάποιο συντονισμός ευρωπαϊκός, τίποτα δεν θα λειτουργεί στους 27. Εγώ είμαι η για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον 2013-2020 και εδώ υπάρχει έλλειμμα μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Και οι βέλτιστες πρακτικές μεταφορά στα εθνικά δίκαια θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα που θα συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερος λοιπόν συντονισμός μας χρειάζεται και θα πρέπει να πούμε στην Επιτροπή να κάνει μια μελέτη για να μελετήσει πώς έχει για όλα τα ευρωπαϊκά θέματα η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Επίσης, το θέμα της ε, επικουρικότητας είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσετε και πρέπει να συνεχίσετε τη δουλειά σας κύριε Στόιμπρ για να δείτε καλύτερα τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Και εμείς θα πρέπει να δούμε ποιος κάνει τι, ποιος είναι υπεύθυνο για το τι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Και ακόμη μία φράση. Ε, Μας λέτε ναι. ότι υπάρχει πίεση πίεση και οι πολίτες αισθάνονται ώρες ώρες ότι κάτι τους καταπνίγει. Αναφέρατε κάποιους αριθμούς, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σημαντικοί οι αριθμοί. Αυτό το οποίο πρέπει να πω όμως είναι ότι οι ρυθμίσεις, οι κανονισμοί, οι οδηγίες, ό,τι κάνουμε, κυρίως αφορούν τον ε, Γεωργία. Έτσι αρχίζουν τα πράγματα. Από εκεί έπρεπε να περάσει κανείς καταρχάς για να προχωρήσει. Αλλά τα πράγματα έγιναν πολύπλοκα και πρέπει να σας πω ότι πρέπει να επικεντρωθείτε στην επικοινωνία και στη σωστή ενημέρωση. Έχετε 30 χρόνια καθυστέρηση για να καταλάβουν οι πολίτες τι ακριβώς γίνεται. Διότι όταν οι πολίτες πλέον στην Ευρώπη δεν καταλαβαίνουν τι λένε, το γραφειοκρατικό τέρας των Βρυξελών ξαναχτύπησε. Και εμείς τι κοστίζουμε εδώ. Το 6% κοινοτικού Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μηχανάκι το οποίο δίνει χρήματα από εδώ και από εκεί. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε με την κοινοτική νομοθεσία είναι να δημιουργήσουμε μία ε, υπεραξία ώστε όλα αυτά να είναι ωφέλη, που κάνουμε εδώ να είναι ωφέλιμα στο σύνολό τους. Ευχαριστώ. Ακούστε, έχουμε 90.000 οδηγίες, κανονισμούς, νομοθετικές πράξεις, ό,τι θέλετε, στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δουλειά έχει γίνει. Η κυρία Λίντα Μακ Ιβεν έχει το λόγο που είναι η συγγήτρια εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Έχει το λόγο Λίντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Σήμερα κάποιο μου είπε ότι χθε στη γερμανική τηλεόραση ένα υπουργό παραπονέθηκε για την ε, νομοθεσία που αφορά την ε, σήμανση στα διάφορα προϊόντα. Και λέει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω να ήρθε κανείς να μας το ζητήσει αυτό. Αντιθέτως, ε, μας ζήτησαν ιδιαίτερως από κάποιες κυβερνήσεις κάποιες να λέει σταματήσουμε την, με το πρόβλημα αυτό της ετικεδοθεσίας λεπτομερού στα διάφορα είδη διατροφής. Τώρα του θέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι εφημερίδες λένε ότι οι Βρυξέλλες επιβάλλουν νομοθεσία, οδηγίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ε, από... Ε, υψηλό επίπεδο επιβάλλονται κάποια τρέπατα. Και οι υπουργοί ήταν αυτοί οι οποίοι αποδυνάμωσαν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φωνά την ετικετοθεσία. Τέλος πάντων. Τώρα, τι κάνουμε με το πρόβλημα το οποίο αφορά την εμπορία ρήπων. Και το πρόβλημα είναι διότι το Συμβούλιο επέμεινε ε, ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που επιτρέπονται και τούτο και τ' άλλο. Τώρα, θα πρέπει να ενθυμούμεθα και το είπατε εσείς, ότι η γρεοκραφία του ενός σημαίνει δικαιώματα για κάποιον άλλο. Πριν από δύο χρόνια, κάποιοι μου είπαν ότι όταν ασχολούνται με θέματα εργασιακά, κάνουμε γραφειοκρατία. Κάποιο άλλο εργαζόμενο μου είπε ότι εργάστηκε στην ευκλογική μου περιφέρεια 7 χρόνια σε ένα εργοστάσιο, 7 χρόνια ε, δούλεψε για διαφορετικά άτομα, πήρε διαφορετικούς μισθούς, δεν του πληρώναν την, ε, το οίκα του, δεν του πλήρωναν κανένα επίδομα ανεργίας, δεν του πλήρωναν διακοπές. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η γραφειοκρατία του ενός είναι τα δικαιώματα του άλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ξέρουμε ότι υπάρχει νομοθεσία, είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σωστά και στην δική μου εκλογική περιπέρεια έχουμε άτομα τα οποία δουλεύουν σε βαριές χειρονακρικές ή άλλες δουλειές και κανένας δεν προστατεύει την υγεία τους. Σε όλα αυτά που συμβαίνουν θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Επίσης, μπορεί κανείς να μιλήσει ε, για την ομοθεσία που αφορά τα εμφυτεύματα, άλλα θέματα που αφορούν την ιατρική και την υγεία. Πώς στο παρελθόν πολλοί θέλανε όποιοι έχουν εμφυτεύματα να μπορούν να καταγράφονται σε ένα... Ε, κατάλογο για να ξέρει καθένας ακριβώς τι γίνεται. Και είπανε κάποιοι άλλοι, ε, ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά». Το, θυμάστε πέρσι τι έγινε με το θέμα των, ε, ε της εταιρείας αυτής ε, η οποία στις πλαστικές στήθους και στην αποκατάσταση δημιούργησε το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω ότι Όταν ήμουν ε, στην Επιτροπή Μεταφορών ασχολήθηκαμε με ένα θέμα που βρούσε την κατάρτιση των οδηγών. Έπρεπε να είναι καλύτερα ώστε να αποφεύγονται τα ε, ατυχήματα. Αυτοί όμως που έπρεπε να αλλάξουν περισσότερα πράγματα στην κατάρταση όντως ήταν οι χώρες τις οποίες υπήρχαν ε, τα μικρότερα ατυχήματα οδικά ή άλλα. Η Σουηδία Φερρυπίν. Εκείνοι όμως χρειάστηκε να κάνουν ε, τις μεγαλύτερες αλλαγές αν ήθελαν να μεταφέρουν την κοινοτική οδηγία που αφορούσε κάτι το ενοποιημένο για την κατάρτιση. Και χρειάστηκε να γίνονται τεστ επί τεστ. Άρα πολλοί παραπονέθηκαν και αυτή η νομοθεσία αναγνωρίζω ότι ήταν αρνητική. Πιστεύω τώρα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ξέρει. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση ε, πρέπει να ξέρει αυτό που κάνουμε θα είναι ε, καλύτερο από αυτό που υπάρχει. Αν υπάρχει κάποια καλύτερη πρακτική, τι πρέπει να κάνουμε να την αποδυναμώσουμε και να μην ε, παίρνουμε αποφάσεις διότι κάποιοι αξιωματούχοι στην Κομισιόν καθισμένοι ωραία στα γραφεία τους αποφασίζουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Επίσης θα ήθελα, κοιτώντας τον κύριο Σνέλχαρτ, να πω το εξή. Πριν από κάποια χρόνια όταν η Επιτροπή εξέτασε την νομοθεσία και είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε απλοποίηση και είδαμε τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια στα είδη διατροφής, είπαν ότι ίσως αυτό θα πρέπει να γίνει. Και μετά το Συμβούλιο στο τέλος ήταν ε, αντίθετο προς το οτιδήποτε, δεδομένο ότι ήταν πάρα πολλές χρόνο να αλλάξουν τα πράγματα. Πολλές φορές λοιπόν το πρόβλημα με την δουλειά την οποία κάνουμε είναι ότι, και αυτό είναι επικίνδυνο, ξέροντας ότι έχουμε χίλιες και τόσες χιλιάδες ε, ε, νόμους, ε, είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλούς το να κάνουν σχόλια. Όταν λένε όμως για να μην ξαγυρίσουμε στην ίδια κατάσταση, ας αλλάξει, αρχίζει το άλλο τραγουδάκι. Όχι, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα. Μία ερώτηση τώρα. Ποιος είναι στην Επιτροπή σας. Έχω ενημέρωση για τι ακριβώς κάνετε. Πόσο εκπροσωπείται η κάθε κοινωνία μεταξύ των μελών σας. Εσείς είστε πολιτικός και δεν λαμβάνετε μόνο υπόψη και την, μόνο τη γραφειοκρατία Φερρυπίν στη βιομηχανία. Πρέπει να εκπροσωπείτε και τους πολίτες. Γι' αυτό, ποια είναι τα μέλη της Επιτροπής σας. Πώς ξέρουμε ότι ο από αυτούς στον τομέα του ε, δεν κάνει λόμπι, δεν υφίσταται πιέση από το λόμπι. Διότι όλα τα πράγματα έχουν δύο απόψεις. Διότι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την κοινοτική νομοθεσία είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν κάποια πράγματα να μην αλλάξουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ιάννα Ρόσμπαχ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Στόιμπερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Είναι πραγματική ευχαρίστηση για μα να μπορούμε να, να συζητούμε μαζί σα Πραγματικά εντυπωσιακά είναι τα ποσά αυτά τα οποία έχετε καταφέρει να εξοικονομήσετε μέχρι στιγμής. Ωστόσο, διερωτάμε για κάτι. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα αυτό το οποίο θα αναπληρωθεί στα τέλη του έτους. Επομένως, ε, προβλέπονται κάποια μελλοντικά προγράμματα για τα επόμενα χρόνια. Είναι εξίσου φιλόδοξα τα προγράμματα αυτά. Πώς θα καταφέρετε να εξοικονομήσετε ένα αντίστοιχο μεγάλο ποσό τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Κρίστα Κλάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στόιμπερ που ήρθατε σήμερα σε εμά. Η συζήτηση ε, δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσα αλλά είναι έτσι και λίγο προκλητική. Ε, εδώ καλούμεθα να αποδώσουμε ευθύνε. Και αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα ενδιαφέρει πολύ του πολίτε. Εγώ εκτιμώ τη δουλειά σα. Ε, εκτιμώ το πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση. Πάρα πολλά από αυτά που είπατε είχαν αποτέλεσμα και νομίζω αυτό πέρασε το μήνυμα. Πράγματι όλοι βρίζουν τις Βρυξέλλες και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Συμφωνώ εδώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Ζήμπα. Ε, θα πρέπει λιγάκι να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο επικοινωνίας ε, και στο μέλλον αυτό να περνάει και καλύτερα στους πολίτες. Και μετά να μιλήσουμε επί της ουσίας. Ο κύριος Γκούτε, ο πρόεδρος, είπε ότι στο περιβάλλον μπορούν να προκύψουν 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Τότε θα πρέπει να διερωτηθούμε και ε, πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας ε, επιβαρύνονται με γραφειοκρατικές ε, διαδικασίες. Αυτό που μου άρεσε πολύ καλά η κυρία Στόιμπα είναι αυτό που είπατε ότι υπάρχουν αίτια διαφορετικής φύσεως, οικονομικά, πολιτικά και εγώ απευθύνομαι τώρα και στους συναδέλφους μου και θέλω να τους πω μερικές φορές και σε πολιτικό επίπεδο δεν φτάνουμε στο διατάφτα. Τι θέλουμε, και τι τελικά αιτήματα υποβάλλουμε. Εχθές, ας πούμε, ψηφίσαμε για το Λούλου ΣΕΕΦ και αυτό υποτίθεται ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα. Ε, εγώ που είμαι γεωργός ε, πρέπει να σου πω ότι μου σηκώνονται οι τρίχες και σκέφτομαι, θα μου, τι θα γίνει τώρα με τη γραφειοκρατία. Το αποτέλεσμα ε, θα πρέπει λοιπόν να είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό και λέω ότι η πολιτική συζήτηση δεν έχει ε, ολοκληρωθεί και όλοι μας ε, πολύ εύκολα κατηγορούμε άλλους. Βεβαίως έτσι χαλαρά προτείνουμε σε αυτούς τους κανονισμούς και τις διατάξεις ότι ναι δεν πρέπει να προκύψει περαιτέρω γραφειοκρατικό άκτος. Και τίτε το ερώτημα, μα βοηθάει αυτό έχετε εσείς ε, καταλήξει, έχετε δει τι βοηθάει αυτό όταν αναφέρεται στις διατάξεις ότι δεν επιθυμούμε να υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία. Και άλλη μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, εγώ έγραψα και θέλησα να σας ρωτήσω ε, τι γίνεται τελικά με την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσει κανείς αυτό. Μπορεί κανείς να πάρει μια οδηγία στη Γεωργία ή οπουδήποτε αλλού, η οποία θα δούμε ότι στη Βαυαρία, παραδείγματος χάρη, εφαρμόζεται τελείως διαφορετικά από ότι στην Ιταλία, ας πούμε. Ε, και τίθε και το ερώτημα, είναι καλύτερα κανονισμός ή οδηγία. Εμείς προτιμούμε τον κανονισμό, γιατί ο κανονισμός εφαρμόζεται πιο εύκολα σε εθνικό επίπεδο. Από την πλούσια εμπειρία που έχετε συλλέξει, ίσως μπορείτε και από αυτού να μας δώσετε κάποιες πρωτοβουλίες. Ε, και τελικά βλέπετε το θέμα της ε, καμπύλης του αγκουριού που μας ε, παιδεύει ε, χρόνια αυτοί που μας έβριζαν τελικά είδατε τι έγινε αυτοί τον ήθελαν τον κανονισμό γι' αυτό βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος των πρώτων ερωτήσεων και τώρα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στις ε, ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ξεκινάμε με αυτά που είπε ο κύριος Γιολάινεν. Λόγω της εμπειρίας που έχω με την εκτελεστική εξουσία, προσφέρθηκα να βοηθήσω. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Περί αυτού πρόκειται. Το γεγονός ότι αυτό βγήκε στη δημοσιότητα είναι, οφείλεται στο ότι εγώ είμαι ο σχετικά μοναδικός γνωστός πολιτικός. Οι υπόλοιποι είναι εμπειρογνώμονες. Ας πούμε από τη Μεγάλη Βρετανία, κυρία Εύαν, σε εσάς απευθύνομαι, έχουμε τον Μάικλ Γκίμπονς από το Λονδίνο, που είναι πρόεδρος της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής ε, της Μεγάλης Βρετανίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος στη Μεγάλη Βρετανία ε, αγωνίζεται για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Στη Γερμανία έχουμε τον κύριο Λούντιβικ, ο οποίος ε, είναι ο πρόεδρος του αντίστοιχου φορέα ελέγχου τυποποίησης. Έχουμε και τον πρόεδρο της Άκταλ, αυτό είναι το είναι Ολλανδικός φορέας. Έχουμε και τον Σουηδό κύριο Πάλμ από τη Στοκχόλμη, ο οποίος ε, προείσταται της ε, Σουηδικής ομάδας. Και να πω κάτι που ίσως είναι σημαντικό για σας. Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, πέντε χώρες από τις 27, οι οποίες έχουν την πολυτέλεια να διαθέτουν ανεξάρτητο φορέα αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες και πριν κατατεθεί νομοσχέδιο, αυτοί οι φορείς έχουν το δικαίωμα κατάθεσης αρνησικήριας Στην Ολλανδία, ας πούμε, η Άκταλ, ο κύριος Ρούτελ, βλέπει ένα νόμο που θα προκαλέσει γραφειοκρατία. Αυτό το θέμα εξετάζεται από την Άκταλ, που είναι ο φορέας ελέγχου, και αν πει ε, ο φορέας καλός ο νόμος αλλά θα προκαλέσει τεράστια γραφειοκρατία, εμείς ε, προτείνουμε να μην ε, θεσπιστεί ο νόμος αυτός και στη Γερμανία η καγκελάριος δεν μπορεί να περάσει νομοσχέδιο αν δεν τον εγκρίνει ο αυτός ο γερμανός, γερμανικός φορές και στην Τσεχία είναι έτσι και στην Μεγάλη Βρετανία. Σε όλες τις άλλες ε, χώρες υπάρχουν φορείς, αλλά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα του βέτο. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα, αλλά κατ' ουσίαν ε, όλοι αυτοί είναι εμπειρογνώμονες και το γεγονός ότι εγώ βέβαια είμαι πρόεδρος αυτό τραβάει έτσι την κοινή γνώμη. Γιατί αν ήμουν ας πούμε καθηγητής ε, οικονομίας από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου ή της Λίλ εντάξει καλή δουλειά θα έκανα αλλά ίσως κανείς δεν θα την πρόσεχε αν θέλετε αυτά ε, που γίνεται τώρα οφείλονται στο ότι σε μεγάλο βαθμό εγώ είμαι γνωστός. Κοιτάξτε, εγώ δεν δυσφημώ τις Βρυξέλλες. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι οι άνθρωποι καταρχήν να συνειδητοποιήσουν πόσο εκτεταμένες είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Λάινεν, ας αφήσουμε το ευρώ. Στη Γερμανία κανείς δεν αναφέρεται ε, σε ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πότε παρουσιάζεται μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ειδήσει, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, σε αντίθεση με ειδήσει από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, στην Αυστρία, ας πούμε, γίνονται πολύ περισσότερες συζητήσεις ε, για τη Βιέννη παρά για τις Βρυξέλλες. Η εντύπωση λοιπόν που προκαλείται στους ανθρώπους είναι ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν πια και τόσες πολλές αρμοδιότητες και με τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει απλά θέλω να καταδείξω πόσο σημαντικές είναι οι Βρυξέλλες για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων ας πούμε στον τομέα των τροφίμων ή των αποβλήτων της προστασίας του περιβάλλοντος αυτό είναι δηλαδή ο στόχος μου, το να προκαλέσω λίγο περισσότερο την κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Βέβαια με την κρίση του ευρώ η κατάσταση έχει αλλάξει. Εχθές η κυρία ε, Μέρκελ επισκέφτηκε του συναδέλφου στην Αθήνα. Παλαιότερα αυτό εμφανίζεται ως αστερίσκος στις εφημερίδες και σήμερα αποτελεί πηχαίους τίτλους. Ε, ίσως και αυτό να μην είναι αρνητικό. Γιατί να αισθάνεται κανείς την Ευρώπη περισσότερο σε ένα φορέα ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση ενοποίησης και πολύ συχνά ε, εθνικά θέματα δεν προβάλλονται. Πρέπει λοιπόν κανείς να διερωτηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητο να υπάρχουν υπερεθνικές ρυθμίσεις. Και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Και εσείς ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό. Για λόγους ασφάλειας ε, μεταφορών είναι καλό που έχουμε ε, ρυθμίσεις για την διάρκεια οδήγησης, ανάπαυσης και όλα αυτά παλιά ήταν καταστροφικά. Ρυθμίστηκαν λοιπόν τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, οι παραδοσιακοί ταχογράφοι αντικαταστάθηκαν από ψηφιακούς ε, ταχογράφους, όπου ο ταχογράφος αναφέρει πόση ώρα οδηγεί ο οδηγός, αν ξεκουράζεται. Τώρα όμως ειδικά στην Αυστρία, για σας το λέω, έχουμε φτάσει στο μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μια φορά ή το πολύ δυο φορές το μήνα να εξυπηρετούν ένα πελάτη και πάνε 8 χιλιόμετρα, αυτούς να τους σταματάνε στον αυτοκινητόδρομο και να σου λένε πού είναι ο ψηφιακός σας ταχογράφος. Και λέει ο άνθρωπος, μα τρελαθήκατε. Ο αστυνομικό το απαντάει, λυπάμαι, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, η Ευρώπη το ζητάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη συνέχεια. Άρα με αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία σε εθνικό επίπεδο που δεν υπάρχει. Για να γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ε, περνάνε κάποια θέματα ως εξαιρέσεις και αυτό είναι δύσκολο. Έχω ενημερωθεί και ξέρω ότι 7 χρόνια πρέπει να περάσουν μέχρι μια οδηγία να αλλάξει οτιδήποτε σε εθνικό επίπεδο. Ο κύριος Βέλε, όχι, ο κύριος Βέλε, ο γενικός σας διευθυντής μου ανέφερε αυτό το στοιχείο ότι οι διαδικασίες είναι τόσο χρονοβόρες. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι η Ευρώπη είναι σημαντική που δεν πρέπει κανείς να τη βλέπει μόνο αρνητικά αλλά και θετικά και πρέπει να σας πω ότι δεν έχω αλλάξει άποψη. Εγώ μην με κατηγορείτε ότι αλλαξοπίστησα, πάντα τα πίστευα αυτά. Και με συγχωρείτε, ε, ποιος οικοδόμησε την Ευρώπη, η δική μας η γενιά. Αν δεν ήμασταν εμείς, η Ευρώπη δεν θα υπήρχε όσοι υπάρχει σήμερα. Το γεγονός ότι η αρχή της επικουρικότητας ε, θα έπρεπε να επικρατεί περισσότερο, δυστυχώς δεν το συζητάνε αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει καμία κυβέρνηση η οποία να λέει ε, τι πρέπει να επαναφερθεί σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένες προτάσεις δεν υπάρχουν. Εγώ έχω 30 σημεία όπου τους λέω κοιτάξτε αυτά να τα ρυθμίσετε σε εθνικό επίπεδο, αυτά περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή η συζήτηση είναι απαραίτητη γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης δεν θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αν δεν υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στην Ευρώπη. Αν όμως το θέλετε αυτό, τότε στην πολιτική συζήτηση πρέπει να υπάρχει και μια συζήτηση για το πού ακριβώς μπορεί να επικρατήσει περισσότερο η αρχή της επικουρικότητας. Να σας πω και κάτι άλλο, για να καταλάβετε τα ποσά. 41 δις ευρώ είναι η πρόταση και από αυτά 100 εκατομμύρια αφορούν εξοικονόμηση στον τομέα του περιβάλλοντος. Στη δική μου την ομάδα με τον Τζον Χοντελες, ο οποίος εκπροσωπεί τις ενώσεις Περιβαλλοντολόγων και ο κύριος Μάρη και αυτός εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών Έρχονται λοιπόν ο Χόντελες και ο και λένε δεν πρέπει να ε, στραγγαλίσετε το περιβάλλον και την προστασία του καταναλωτή. Ας πούμε υπάρχει μια πολύ σημαντική πρόταση η οποία είναι επιτέλους οι υπολογισμοί του φόρου κύκλου εργασιών να γίνονται ηλεκτρονικά. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν. Δηλαδή Παρότι αυξάνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι επιχειρήσεις ήταν αναγκασμένες να αναφέρουν τον κύκλο εργασιών σε χαρτί. 7 ευρώ κόστιζε αυτό. Ηλεκτρονικά όμως 1 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Αυτό θα αποτελούσε ελάφρυνση για τα 23 εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα σήμαινε 18 δις ευρώ εξοικονόμηση. Μόνο που πολλές χώρες δεν το χρησιμοποιούν αυτό. Στη Γερμανία ναι. Και στη Γερμανία εξοικονομούν 4 δις ευρώ. Και θα το ελέγξουμε λιγάκι να δούμε ποιος δεν το κάνει πια. Αυτά ας πούμε είναι θέματα όπου μπορεί κανείς να πει η Ευρώπη κάτι κατάφερε. Ή άλλο παράδειγμα. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών. Γιατί να ισχύει και για τις ε, μικρού, μικρότατες επιχειρήσεις που αυτές δεν έχουν διεθνείς ε, εμπορικές ανταλλαγές, εξυπηρετούν μόνο σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Στο κοινοβούλιο σας το συζητήσατε αυτό δύο ολόκληρα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτή συζήτησε το θέμα για άλλα δύο-τρία χρόνια, μετά το Κοινοβούλιο άλλα δύο, μετά το Συμβούλιο άλλα δύο, φτάσαμε στα 7 χρόνια και εμένα μου επιτίθενται και μου λένε εσύ το ζήτησες το 2007, φτάσαμε στο 12 και τίποτα δεν έγινε. Και εκεί μας αμφισβητούν όλες, όλους. Θέλω λοιπόν να σας δείξω πού είναι τα πιο προφανή παραδείγματα, όχι στο περιβάλλον στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της αγοράς εργασίας και κυρίως στο εταιρικό δίκαιο. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, αλλά αυτή είναι μια πρόταση της τάξης των 18 ε, δις ευρώ που νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόταση. Κυρία Ρόσμπαχ, εγώ προσπάθησα να παρουσιάσω παραδείγματα και συγκεκριμένα ποσά. Και θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιο ισχυρή ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Δηλαδή, όταν ας πούμε το κοινοβούλιο μιλάει για τους λαμπτήρες, τους οικονομικούς λαμπτήρες, κανείς δεν το κατάλαβε, κανείς δεν το συνειδητοποίησε. Μετά, ελήφθη μια απόφαση και από το κοινοβούλιο και μετά έξανε κατά την εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιθυμώ η διαδικασία πολιτικών αποφάσεων αυτή η διαδικασία να γίνεται περισσότερο σε εθνικό επίπεδο. Κύριε Λάνεν, εγώ τσακώθηκα με τις εφημερίδες. Μέχρι πριν από δύο χρόνια η εφημερίδα Bild, παρότι γράφει πολλά για την Ευρώπη, η Bild δεν έχει εδώ στις Βρυξέλλες ανταποκριτή. Ή ας πάμε στη Γερμανία. Το Spiegel, που είναι ένα από τα σημαντικότερα, καλύτερα περιοδικά ε, στην Ευρώπη από τα πιο έγκυρα. Το Σπίγκελ έχει 50 συντάκτες στο Βερολίνο, ε, αλλά εδώ στις Βρυξέλλες είχε μόνο ένα και έφερε τώρα πρόσφατα και άλλον ένα, έχει δύο. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι σωστή η ενημέρωση που γίνεται για τη δική σας τη δουλειά σε σχέση με τα εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια. Αυτό είναι εκείνο που με απασχολεί και γι' αυτό τους λέω, μα ξέρετε πόσες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις ε, που σας επηρεάζουν προέρχονται από την Ευρώπη. Δεν είναι ότι θέλω να ε, δυσφημίσω την Ευρώπη, αλλά ξαφνικά οι άνθρωποι ξυπνάνε και λένε πώς γίνεται το, τι γίνεται εδώ. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να συμβάλλω έτσι ώστε τα εθνικά ε, κοινοβούλια και τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις Βρυξέλλες. Βέβαια όλα αυτά τώρα τα επισκιάζει η συζήτηση για το ευρώ. Και να κάνω και άλλη μια παρατήρηση. Ο Jean-Claude Juncker, κολλητός μου, πολύ καλός μου φίλος, το 99, πριν από αρκετό καιρό δηλαδή, ήδη το 99, έδωσε έτσι μια πολύ σημαντική συνέντευξη στο περιοδικό Spiegel και εκεί είπε σχεδόν κατά λέξη αυτή είναι η Ευρώπη των ελίτ. Θα δείτε τώρα τι θα πω. Είπε λοιπόν περίπου. Κοιτάξτε, είπε λοιπόν και παραθέτω. Αποφασίζουμε κάτι στην Ευρώπη, μετά περιμένουμε τι αντιδράσεις, που όμως δεν υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι αποφασίσαμε και εμεί συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Αυτά είπε ο κύριο Γιούγκερ. Πολύ συχνά λοιπόν έτσι ελήφθησαν οι αποφάσεις. Και σήμερα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο τη συμμετοχή των ε, πολιτών σε αυτή την ευρωπαϊκή διαδικασία. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε ένα μεγάλο εγχείρημα η Ευρώπη δηλαδή δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτά που καλείται να υλοποιήσει. Και το λέω αυτό σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που βλέπω τι ακριβώς διαδραματίζεται. Άρα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας γιατί τόσο οι μικρές όσο και οι αποκαλούμενες ε, μεγάλες χώρες, ε, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, μόνοι μας και οι μεγάλοι δεν θα έχουμε τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε από ότι όταν εμφανιζόμαστε ως ε, Ευρωπαίοι και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ωφελεί και την Αυστρία, το Τυρόλο, τη Βαβαρία, την Αλσατία, ε, τη Γαλλία, το Έσεξ, τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα, τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, και αυτό θα το κάνουμε του χρόνου, θέλω να υπάρχει ένα είδος διαθήκης. Η νέα επιτροπή το 2014 θα πρέπει να συστήσει κάτι σαν την Άκταλ στην Ολλανδία ή το Ρέγγελράντε στη Σουηδία ή αυτή η επιτροπή που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία να έχουν ομάδες επαϊόντων έτσι ώστε τα θέματα της γραφειοκρατίας να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα και μάλιστα και σε αντιπαράθεση με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, ίσως να βάλαμε το πρώτο λιθαράκι ε, και η συνέχεια να υπάρξει κατά την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά μου και πρέπει να σας πω ότι σκοπεύω και να τσακωθώ και με τις εθνικές διοικήσεις. Θα πάω ε, στα διάφορα κράτη-μέλη, θα θέσω το δάκτυλο στον τύπο των ύλων και θα τους πω αυτό στυλιτεύω, για δέστε πώς γίνονται τα πράγματα στη Φινλανδία, λιγότερη γραφειοκρατία, πολύ πιο ανοιχτά και εσείς εδώ στη χή χώρα ας πούμε ε, έχετε συντάξει 30 σελίδες για το ίδιο πράγμα. Βεβαίως και γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, εφαρμοστικές ρυθμίσεις. Ε, σε κάποιες χώρες αυτές ε, είναι δύο σελίδες και σε άλλες 30. Προφανώς και υπάρχουν διαφορές. Βεβαίως και κυρία Κλάς, οι Βρυξέλλες, μήπως είναι καλύτερα οι οδηγίες να θεσπίζονται επιτόπου, γιατί θα έχουμε απλά μία ενιαία νομοθετική βάση, αλλά όχι διαφορετικούς νόμους. Γιατί όταν εφαρμόζεται μια οδηγία μέσα από ένα νόμο, ε, κατ' ουσίαν προσθέτουμε ε, τη δική μας ε, την ερμηνεία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αφήνει κανείς ένα περιθώριο ερμηνεία στα κράτη-μέλη. Όμως, κυρία Κλάς, αυτή η ερμηνεία, κατά τη δική μου την άποψη, και εδώ πάω πάλι πίσω, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες αρμοδιότητες και ελέγχους. Η Κομισιόν πρέπει να μπορεί να πει αυτό που κάνεις εσύ, χι χώρα, δεν γίνεται. Ε, εδώ είσαι αντίθετος με αυτά που θέλουμε εμείς, που θέλουμε να ενοποιήσουμε την Ευρώπη. Και μέχρι τώρα η Γενική Γραμματεία είπε ότι θα δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε τις διατάξεις. Θα θέλαμε λοιπόν να μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη εναρμόνιση ώστε όλες οι οδηγίες μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο με καλύτερο τρόπο. Και έτσι η δημιουργούμενη γραφειοκρατία από τις εθνικές διοικήσεις να μειωθεί. Τι θέλουμε τελικά να έχουμε. Να λένε οι άνθρωποι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θεσμικά όργανα, αλλά κυρίω η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατάλαβαν ότι υπάρχει πρόβλημα διοικητικού άχθους και όντως θα πρέπει, εφόσον υπάρχει πρόβλημα, να προσπαθήσουμε να το βρούμε μια λύση. Βεβαίω θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα. Και όπως σας είπα, για την προστασία των καταναλωτών, οι προτάσεις μείωσης αφορούν 200 εκατομμύρια και για προσθέτει περιβάλλοντος 100. Διότι κάθε φορά που μειώνεται μείωση, πάντα προσπαθούμε να δούμε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την πραγματική προσοχή του περιβάλλοντος. Η δική μας η προσέγγιση σε αυτήν την περίπτωση ήταν πάρα πολύ προσεκτική και διότι και ο εκπρόσωπος της προσίας των καταναλωτών ήταν εντελ... κάθετα αντίθετος με την ε, γραμμή αυτή. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Ιρλανδός συνάδελφος. Στον οποίο αρέσουν όλες αυτές τις συζητήσεις, αλλά πολλές φορές βάζει τροχοπέδι. Προσπαθεί όχι μόνο να μειώσει τη γραφειοκρατία, αλλά να δει και ποια είναι οι επιπτώσεις της κάθε πράξης. Διότι μπορεί να μειώσεις κάτι από τη μια και να αποδυναμώσεις το σύστημα από την άλλη. Όπως σας είπα λοιπόν και προηγουμένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να βρούμε τη χρυσή τομή μέχρι το να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς ε, καμία ρύθμιση ή να ρυθμίσουμε τα πάντα. Και κάθε κράτος, οι πολιτικοί που εκπροσωπούν το κράτος, όπως ξέρετε, δεν έχουν και πολύ καλή μέλη. Αλλά υπάρχουν ε, κράτη, δημόσιες διοικήσεις όπως ε, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία που οι πολίτες εμπιστεύονται το κράτος. Και πιστεύουν ότι πρέπει το κράτος να ρυθμίζει τα πάντα για να λειτουργούν σωστά. Εγώ προσπάθησα να κάνω συζήτηση εδώ να πω κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως δεν μπορώ να τα πω όταν γίνεται η γιορτή της μπύρας τον Οκτώβριο. Δεν είναι το κατάλληλο επίπεδο. Εδώ όμως επειδή είστε πολιτικοί σας λέγω κάποια πράγματα και επαναλαμβάνω υπάρχει όντως έλλειμμα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες τι κάνει η Ευρώπη, για ποιο λόγο και γιατί καλύτερα κάποια πράγματα που κάνει η Ευρώπη να συνεχίσει να τα κάνει. Αλλά βεβαίως υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας. Αυτά ήθελα να πω. Μ' ακούσατε αρκετή ώρα. Τώρα κλείνω το στόμα μου και σας ακούω. Okay. Bis um halb eins. Also da können wir die Kollegen, die sich noch gemeldet haben, ich bitte äh, noch dran nehmen. Und ich würde doch bitten, Ήθελα να δώσω το λόγο συναδέλφου που δεν έλαβαν ακόμη το λόγο. Δύο λεπτά όμω ο καθένα παρακαλώ για να μπορέσουν όλοι να μιλήσουν. Καρ Σλούτερ. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα αν θέσετε ως προϋπόθεση το γεγονός ότι ε, η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου θα οδηγήσει σε χαμηλότερα πρότυπα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχαμε μια συγκεκριμένη νομοθεσία για την ποιότητα των τροφίμων, μα είχαν πει κάποιοι, οι οποίοι φτιάχνανε gingerbread για παράδειγμα στην Αγγλία, ότι δεν υπάρχει λόγο να δημιουργηθούν κανονισμοί για τα πάντα, αλλά θα πρέπει να προβλέπονται για συγκεκριμένα προϊόντα πολλέ εξαιρέσει. Το πρόβλημα είναι ότι αν έχουμε πολλέ εξαιρέσει, τότε ε, δημιουργείται ένα πρόβλημα, δημιουργείται περισσότερο διοικητικό άχθος. Αν για παράδειγμα για το ψωμί ή το κέντζερ πρέπει να υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε εξαιρέσει, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να προβλέπονται και πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Νομίζω ότι πολλέ φορέ η γραφειοκρατία τελικά προέρχεται από το μέλημα ορισμένων επιχειρήσεων να εξαιρεθούν από κάποιου κοινοτικού κανονισμού. Οι επιχειρήσει τελικά είναι αυτέ οι οποίε δημιουργούν περισσότερο διοικητικό φόρτο πολλέ φορέ. Θα ήθελα επίση να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το ζήτημα τη αρχής επικουρικότητας, που τελικά η επικουρικότητα ισχύει και που όχι. Και κάτι ακόμα. Βλέπω ότι έχουμε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπονται τα πάντα από την αρχή. Ουσιαστικά προκειμένου να επιτραπεί κάτι, να ισχύει κάτι νομικά, θα έπρεπε να υπάρχει και ένας νόμος γι' αυτό. Νομίζω ότι εναλλακτικά θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ένα άλλο μοντέλο. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάνταρτ, κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. Αν όμω μετά μια χώρα θέλει να προχωρήσει με μια δική τη εξειδικευμένη νομοθεσία, τότε α αντιστρέψουμε το βάρο τη απόδειξη. Να τους πούμε δηλαδή, μπορείτε εσείς στη χώρα σας να κάνετε αυτό το οποίο θέλετε, αν όμως δούμε τελικά ότι προωθείτε μόνο τη δική σας βιομηχανία και, και, και ότι για αυτό το λόγο ουσιαστικά θέλετε να έχετε μια εξειδικευμένη νομοθεσία, τότε να μην το επιτρέψουμε. Αν όμω μια χώρα θέλει να έχει μια δικιά τη εξειδικευμένη νομοθεσία προκειμένου να προστατεύσει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, τότε θα πρέπει να μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο, θα λειτουργεί πολύ πιο καλά εσωτερική αγορά και δεν θα έχουμε τόσο κεντρικό χαρακτήρα στην νομοθεσία και στου κανονισμού. Entschuldigung, habe ich nicht gehört. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Στόιμπερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης να βλέπουμε τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική εφαρμογή των όσων συζητάμε και αποφασίζουμε. Καταρχάς, αυτό πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς νομοθετούμε, για ποια θέματα και πώς οι νομοθεσίες αυτές μεταφέρονται μετά στα κράτη-μέλη. Να βλέπουμε επίσης ποιες είναι οι συνθήκες ανταγωνιστικότητας οι οποίες ισχύουν, πώς επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα από τις νομοθεσίες μας. Και το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να έχουμε μια κεντρική νομοθεσία που δεν θα χρησιμοποιείται όμως από τα κράτη-μέλη προκειμένου να γίνονται πιο ανταγωνιστικά από κάποια άλλα κράτη-μέλη. Η Λίντα Μακαΐβαν αναφέρθηκε σε αυτό πριν από λίγο. Οι κανονισμοί πολλές φορές είναι καλύτεροι από τις οδηγίες, γιατί ακριβώς η μεταφορά είναι πιο άμεση και καλύτερη. Και στα πλαίσια των κανονισμών πολλές φορές προβλέπεται ένα μεγάλο περιθώριο ευελιξίας. Κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μην βαρύνουμε ιδιαίτερα κάποιες μικρές και μεσές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ενδεχομένω μια μεγαλύτερη ευελιξία. Βλέπουμε βέβαια πώς αντιδρά και ο κόσμος, η κοινή γνώμη, οι επιχειρηματίες. Μας είπατε για αντιδράσεις στη Γερμανία, έντονες αρνητικές. Από την άλλη βλέπουμε ότι στην Αυστρία υπάρχουν πολλοί που είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την κοινοτική νομοθεσία. Μήπως τελικά δεν έχει να κάνει με την νομοθεσία αυτή καθ' αυτή, αλλά με την εφαρμογή της κοινοτική νομοθεσίας. Οι αποδοκιμασίες, οι επιδοκιμασίες τελικά έχουν να κάνουν με την εφαρμογή επιτόπου και όχι τόσο με την ουσία της νομοθεσίας. Ας δούμε δηλαδή πώς εφαρμόζονται επιτόπου σε εθνικό επίπεδο όλες αυτές οι ρυθμιστικές διατάξεις. Αυτό θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε αν τελικά η εθνική μεταφορά είναι εξίσου σαφής και συγκεκριμένη όσο ήλπιζε αρχικά η κοινοτική νομοθεσία ότι θα έπρεπε να είναι. Ας εξετάσουμε λοιπόν εκ του σύνεγγης περισσότερο την εθνική μεταφορά και την επιτόπου εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων. Νομίζω ότι είναι λογικό να κάνουμε κάποια λάθη, να σφάλουμε που και που. Λυπάμαι ενδεχομένω για κάποια πράγματα που είπα πριν από λίγο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ε, δεν λειτουργεί πάντως, πάντα κανείς με τον ίδιο τρόπο όταν λειτουργεί στη χώρα του, όταν είναι εθνικός βουλευτής. Πολλές φορές η οπτική γωνία είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πάντως πάρα πολύ θετικό το ότι μας δίνεται δυνατότητα να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σήμερα εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως ανάλογη συζήτηση να γίνει και στα κράτη-μέλη, μόνο ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Μέρκελς. Σας ευχαριστώ κύριε Στόιμπερ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επισκόπηση της κατάστασης. Θα ήθελα να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι δεν έχουν επιληθεί, μόλον ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις. Και εσείς ο ίδιος είπατε ότι εκκρεμούν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Πρώτον, αν αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγίων, οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν είναι τόσο δύσκολη η επιτόπου εφαρμογή του, αν η εφαρμογή του οδηγεί σε τόσο μεγάλη απόκληση από το ένα κράτο μέλο στο άλλο, μήπω θα έπρεπε οι οδηγίε αυτέ απλώ να γίνουν κανονισμοί, μήπω θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε τελικά την πληθώρα των οδηγιών και να πηγαίνουμε ευθύ αμέσω σε κανονισμού. Οι κανονισμοί δεν απαιτούν εθνική μεταφορά, θα ήταν ενδεχομένως μια επιλογή βαρέως πυροβολικού που όμως θα μας βοηθούσε να έχουμε πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτόπου. Έπειτα, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είχαμε έναν πιο αποκεντρωμένο χαρακτήρα επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό θα βοηθούσε ενδεχομένω τις μικρομισές επιχειρήσεις. αν υπήρχε δηλαδή και μια εθνική υποστήριξη προς την εφαρμογή των κοινωτικών αποφάσεων. Μας είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν πολλές διαφορές στην ε, εφαρμογή και ότι αυτό οδηγεί τελικά πολλές φορές σε κατασπατάληση πόρων. Δεν θα έπρεπε να προσβλέπουμε σε ένα ελάχιστο επίπεδο εφαρμογής στα κράτη-μέλη, να δίνουμε για παράδειγμα μία προθεσμία 8 ετών προκειμένου μία οδηγία να μπορεί να εφαρμόζεται πλήρως τελικά. Τέταρτη παρατήρηση. Μας είπατε ότι φύστανται πολλά διαφορετικά δεδομένα όσον αφορά την εφαρμογή. Θα ήταν καλύτερα τα δεδομένα αυτά να ήταν πιο ομοιογενή και συγκεκριμένα. Αλλά θα έπρεπε τότε να διευθετήσουμε και κάποια ζητήματα εμπιστευτικότητα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω ακόμα περισσότερο. Η εμπιστευτικότητα, η ιδιωτικότητα θα πρέπει να προστατεύεται. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να είχαμε μία πιο κεντρική προσέγγιση όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη διασύνδεση προκειμένου να καταφέρνουμε να έχουμε αυτές τις πληροφορίες για την εφαρμογή των οδηγιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε έπειτα και στους ελέγχους και είπατε ότι πολλές φορές υπάρχει επικάλυψη στους ελέγχους. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτέ, μη κυβερνητικέ οργανώσει, ακόμα και διεθνεί οργανώσει στο Συμβούλιο τη Ευρώπη που ασχολούνται με τον έλεγχο της ε, Κοινωνική νομοθεσία κατά την επιτόπου εφαρμογή της. Μας είπαν ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο και πόρους στην επικάλυψη. Πάρα πολλοί οργανισμοί κάνουν τα ίδια πράγματα. μήπω δεν θα έπρεπε να βελτιώσουμε και το σύστημα αυτό. Και εφόσον μιλάτε με έναν τόσο ομοσπονδιακό στυλ, μήπω θα έπρεπε να καταλήξουν περισσότερο σε μια ομοσπονδιακή ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Πίτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένοι από εμά περίμεναν δύο ώρες για να θέσουμε τις ερωτήσεις μας. μήπω θα έπρεπε να περιορίσετε λίγο το χρόνο ομιλίας. Ξέρετε, Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, πέρα από τον κύριο Ζίμπερ, που θα μπορούσαν και αυτοί να πάρουν το λόγο για να πούν ορισμένα πράγματα. Κύριε Στόιμπερ, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ επίσης για τα επιτεύγματά σας. Τα όσα πετύχατε όσον αφορά τον περιβαλλοντικό φόρο είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι οι επιτυχίες αυτές, αυτές θα σας οδηγήσουν στο να είστε ακόμα πιο αποτελεσματικός στο έργο σας. Και συμφωνώ με τον κύριο Ζίμπερ ότι υπάρχουν σημεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν, όμως στη Γερμανία να γνωρίζουμε ήδη πάρα πολύ καλά την εργασία την οποία κάνετε. Ξέρετε ότι ε, θα μπορούσαμε ακόμα και να απευθυνθούμε στους ε, ηθήνοντές μας, ακόμα και στην ε, κυρία Μέρκελ, σε μια παλιότερη συνέντευξη τύπου, είχε επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως ότι αν υφίστανται τέλος πάντων τέτοιες αμφιβολίες ή ενδιασμοί θα πρέπει να ασχοληθούμε κάπως με το ζήτημα αυτό. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπε η κυρία Μακέιβεν. Θα μπορούσα να απευθυνθώ επίσης και στον αρμόδιο Γερμανό υπεύθυνο υπουργό να αφορά όλα αυτά τα ζητήματα για την επισήμανση των προϊόντων. Ξέρετε ότι στη Γερμανία πολλές φορές πρέπει να πετυχαίνουμε μια συμφωνία ανάμεσα στις διαφορετικούς, διαφορετικές πολιτικές ομάδες στα πλαίσια του κυβερνητικού συνασπισμού. Το σημαντικό είναι κάθε φορά να καταλήγουμε σε μία προσέγγιση η οποία θα είναι θετική για τους, καταναλωτε... για τους Όσον αφορά τώρα την υγιεινή των τροφίμων, και η κυρία Μακέβα αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Κύριε Στόιμπερ, το δικό σας πολιτικό κόμμα ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό, εξέφρασε κάποιες ιδέες κατά της γραφειοκρατίας Για την ε, ηλεκτρονική τομογραφία επίσης είχαν ε, ληφθεί κάποιες αποφάσεις, ακόμα και στον τομέα αυτό ε, θέλουν να πετύχουν μια ευρωπαϊκή λύση, μια ευθυγράμμιση με μείωση του διοικητικού φόρτου. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι αν δεν καταφέρνουμε τελικά να πετύχουμε ορισμένα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει τουλάχιστον αυτά να γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι ότι κινδυνεύουμε στην Γερμανία να έχουμε υπουργού οι οποίοι θα απορρίψουν ευρωπαϊκές λύσεις, θα καταλήξουμε τελικά με μια νέα κυβέρνηση στο μέλλον, η οποία τελικά θα υιοθετήσει μόνο εθνικές λύσεις, οι οποίες τελικά θα βάλουν κατά της γερμανικής επιχειρηματικότητας. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ που σεβαστήκατε αυτά τα δύο λεπτά. Η Φρανσουάς Γκροστέτ έχει το λόγο. θα ήθελα να σας πω ότι με μεγάλη ευχαρίστηση σας άκουσα. Πρέπει επίσης να πω ότι αυτά που μας είπατε ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτά τα οποία αισθάνονται και οι πολίτες μας και οι συμπολίτες μας. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει πολύ γραφειοκρατή γιατί είναι πληθωρική η δίκηση και έχει μεγάλη βαρύτητα Άρα είναι και ευθύνη των πολιτικών που άφησαν αυτή την διοίκηση να γίνει τόσο επιθαρμία. Αν είχαμε όμως λιγότερη γραφειοκρατία, θα είχαμε λιγότερο άχθος και θα ήταν καλύτερη και επιχειρήση. Αν πιστεύετε ότι η Ευρώπη είναι Ευρώπη των καταναλωτών και ξέχασε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ε, διάφορες επιχειρήσεις της υπόλοιπης είναι γιατί σήμερα διερχόμαστε κρίση και οι επιχειρήσεις ζουν δύσκολα μέσα σε αυτή την κρίση σήμερα. Επίση, υπάρχει το θέμα της ευθύνη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και καθώς και του Συμβουλίου. Όταν δούμε το πρόβλημα του ευρωπαϊκού ε, διπλώματος ευρεσιτεχνίας και όταν δούμε τι έχει γίνει για να καταλήξουμε κάπου δεδομένου ότι μπλοκάρουν κάποια κράτη-μέλη την όλη διαδικασία, τι να πω. Υπάρχει πραγματικά νομική αστάθεια που βαρύνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις μας. Και εμείς ε, έχουμε να υπομισθούμε ένα μέρος της ευθύνη εδώ. Δεν το άκουσα το λένε οι συνάδελφοι, διότι πολύ συχνά εμείς επιδεινώνουμε την κατάσταση, ζητούμε περισσότερη νομοθεσία, Πράγμα το οποίο βαρύνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργεί αστάθεια. Διότι πάντα αναμένουν μια κάποια αναθεώρηση της νομοθεσίας για να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν ε, πάρα πολύ πολύπλοκοι φάκελοι του οποίου πρέπει να παρακολουθήσουμε. Και όταν μας λέτε σήμερα ότι ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι έτοιμος να δημιουργήσει μια νέα γενική διεύθυνση για τι επιπτώσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ανησυχώ. Τι σημαίνει, ακόμη περισσότερη δίκηση. Θα προτιμούσα οι επιπτώσεις να μελετηθούν από κάθε γενική διεύθυνση, αλλά να μην δημιουργήσουμε και μια νέα δομή η οποία θα καπελώσει όλες τις άλλες. Δεν νομίζω ότι μας χρειάζεται κάτι τέτοιο. Καλύτερη νομοθεσία ζητούμε όλοι. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι το θέμα αυτό αναφέρθηκε για πάλους. Λοιπόν, κύριε Στόιμπερ, δεν ζητά κανένας άλλος συνάδελφος το λόγο, σας δίνω το, εσάς το λόγο για να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ. Κύριε Γκρότε, ξέρω ότι καταχράστηκα τις υπομονή σας, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλα πράγματα να εξετάσετε σήμερα, αλλά θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση ήταν ανοιχτή, πολύ καλή ήταν μια συζήτηση η οποία βοηθάει στην ε, συνειδητοποίηση θεμάτων. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σχετικά με τις συνέπειες ε, των ε, νομοθετικών ρυθμίσεων. Και κύριε Σλούτε, εσείς υποβάλλετε μια καθοριστική σημασία ερώτηση ή παρατήρηση. Η μείωση της γραφειοκρατίας δεν σημαίνει απαραίτητα νόθευση των προδιαγραφών. Αυτό θα ήταν λάθος. Ε, το συζητήμε αυτό, ε, παραδείγματο χάρη συζητάμε για την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να του πούμε ότι κοιτάξτε μια μεγάλη επιχείρηση πρέπει να καλύπτει αυτές τις προδιαγραφές και μια μικρή επιχείρηση με ε, πέντε υπαλλήλου αυτή θα έχει έκπτωση στις προδιαγραφές. Δεν γίνεται αυτό, ούτε απέναντι στον καταναλωτή. Οι προδιαγραφές κατ' ουσίαν πρέπει να παραμένουν οι ίδιες. Η μείωση της ε, γραφειοκρατίας δεν πρέπει να οδηγεί στην ε, υπονόμευση ε, των πολιτικών οριζόμενων προδιαγραφών. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα και αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που κάνει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Δηλαδή, πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου για αυτές ειδικά δεν θα ζητούνται ορισμένες γραφειοκρατικές διατάξεις, η εφαρμογή κάποιων διατάξεων. Τώρα λοιπόν τι το εξή το θέμα, κατά πόσον ενδεχομένως θα πρέπει να κατέβει το επίπεδο για όλους ή αν θα πρέπει για μεγάλες επιχειρήσεις να παραμείνει το επίπεδο και να πέσει για κάποιες μικρές. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται και η Κομισιόν του χρόνου θα τοποθετηθεί επ' αυτού. Εάν λοιπόν και εσείς ε, θέλετε να συμμετάσχετε, πάρα πολύ ωραία. Εγώ, ε, βλέποντας ότι μία μεγάλη επιχείρηση, ε, το 1% του κύκλου εργασιών του, το διοχετεύει στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Μία επιχείρηση με πάντο, μεσαία με πάνω από 52 υπαλλήλου το 5% και μια μικρή επιχείρηση ε, είναι αναγκασμένη περίπου το 10% του τζίρου της να το διαθέσει για την τήρηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτά είναι εντυπωσιακά στοιχεία και πρέπει να δουλέψουμε γιατί το μέλλον της Υπήρου μας εξαρτάται από μεγαλύτερες ε, και περισσότερες επιχειρηματικές ε, πρωτοβουλίες. Άρα δηλαδή πολιτικός είναι ο στόχος. Αυτά που είπατε τώρα σχετικά με την επικουρικότητα πραγματικά ε, είναι εντυπωσιακά. Κύριε Σνελχώστ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι επειδή μιλήσετε για την Αυστρία και τη Γερμανία, κοιτάξτε, χρειαζόμαστε όσο έχουμε οδηγίες, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο εθνικών διοικήσεων για θέματα εφαρμογής νομοθετικών ε, διατάξεων. Αυτό το εκφράζουν πολύ ως αίτημα και εγώ το στηρίζω και τους ε, αναφέρω πολλά παραδείγματα, τα 74 αυτά παραδείγματα που έχω συγκεντρώσει. Κυρία Μέρκης, κανονισμοί ή οδηγίες. Ετέθη αυτό το ερώτημα και από την κυρία Γκροστέτ. Ε, και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ε, κανονισμούς. Ε, πράγματι, η τάση είναι προς εκπόνηση περισσότερων κανονισμών. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης, δεν θα πω ονόματα, αλλά προς Ανατολάς, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στην επάρκεια. Ε, δεν ξέρω αν είναι πάντα κακή πρόθεση. Πολλές φορές λείπουν και γνώσεις. Ανεπάρκεια γνώσεων. Άρα δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο διάσκεψης κορυφής. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν περισσότερα για καλύτερη εφαρμογή, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει και ε, μεγαλύτερος έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φτάνω λοιπόν στο κέντρο τεκμηρίωσης όπου θα πρέπει να κατατίθενται κάπως οι οδηγίες για να ξέρει και η Κομισιόν να έχει το γενικό έλεγχο του τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα δηλαδή περισσότερη Ευρώπη και περισσότερος έλεγχος. Κύριε Λίζε, συμφωνώ μαζί σας. Όσον αφορά τις εκπομπές, πράγματι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί σε εθνικό επίπεδο. Ή μάλλον το να ρυθμιστούν οι εκπομπές σε εθνικό επίπεδο θα ήταν παντελώς λανθασμένο. Σήμερα ε, πολλοί λένε ότι πρέπει να ξαναπροβληθεί το θέμα της Ευρώπης. Για μένα η Ευρώπη είναι η απάντηση στους δύο αιματηρούς πολέμους και κυρίως η απάντηση στην ευθύνη των Γερμανών από το δεύτερο πόλεμο. Για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου όλα αυτά βέβαια είναι ιστορία, είναι παρελθόν. Ε, δεν πείθενται πείθονται από τους πολέμους και από την Ευρώπη του 20ου ε, αιώνα. Σήμερα η απάντηση είναι η παγκοσμιοποίηση. Αυτή η Ευρώπη έχει τεράστια προβλήματα. Είμαστε ε, ήπειρος με όλο και λιγότερους ανθρώπους σας. Η Κομισιόν λέει το 2014 η Ευρώπη θα έχει 50 εκατομμύρια λιγότερους κατοίκους ενώ ε, ο παγκόσμιος πληθυσμός το ίδιο χρονικό διάστημα από 7 δις θα πάει στα 9 δις. Υπάρχουν λοιπόν σαφώς λόγοι γιατί χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Κύριε Μέρκης, ε, μιλήσατε για κανονισμό ή επικουρικότητα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή επιτροπή τελική ανάλυση αυτό που δεν προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και αν θέλετε να έχουμε τη δική μου την πολιτική εκτίμηση, το Συμβούλιο τώρα έχει γίνει πιο ισχυρό και η Κομισιόν αποδυναμώθηκε και το Κοινοβούλιο είναι κάπου στη μέση, ανάμεσα στους δύο. Νομίζω λοιπόν ότι η σημασία του Συμβουλίου δεν είναι ικανοποιητική. Παράδειγμα, Όταν ε, συνεδριάζει το Συμβούλιο Κορυφής έχουμε 27 διαφορετικές συνεντεύξεις τύπου. Και τι λέει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ιταλός, ε, η καγκελάριος λένε όλοι εγώ ε, εκπροσώπησα τα ιταλικά συμφέροντα, εγώ περασπίστηκα τη Γερμανία. Ε, το ίδιο όμως λέει και ο Βούλγαρος. Λέει, εμφανίζεται στην έντευξη τύπου και λέει εγώ υπερασπίστηκα με όλο μου το βάρος ε, τα συμφέροντα της Βουλγαρίας έναντι αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως εγώ δεν μπορώ να τα αλλάξω. Εγώ προσπαθώ απλά να το επισημάνω και να εξάγω τα συμπεράσματα. Για την προστασία των δεδομένων, να σας πω το εξής. Όταν αναφέρεται μία ημερομηνία, θα πρέπει αυτό να αρκεί. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον πολίτη να στέλνει τρεις φορές τα στοιχεία του. Μια στο κράτος, μια στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια στην περιφέρεια. Ε, κάποια στιγμή θα πει και ο πολίτης, μα τα έχω στείλει τα στοιχεία μου. Πήγα στη Μεγάλη Βρετανία, θαυμάσιο παράδειγμα και πήγα στον αρμόδιο υπουργό Ρίσκ, ο οποίος υπουργό μου είπε, ε, καταρχήν διαπιστώσαμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν πάνω από 22.000 νομοθετικές διατάξεις. Περισσότερες από αυτές των Ιταλών και δεν ξέρουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Ήδη οι Βρετανοί το είπανε. Η κυβέρνηση Κάμερον, αυτή μας το είπε και μας είπε, διαπιστώσαμε, ότι στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αγγλία μία γελάδα εξετάζεται από 19 διαφορετικούς φορείς για διάφορους λόγους. Και μου είπε, η Αγελάδα χαίρεται βέβαια γιατί είναι ε, στο κέντρο της προσοχής, αλλά δεν χαίρεται ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Γιατί λοιπόν πρέπει η Αγελάδα να εξετάζεται 19 φορές, γιατί να πρέπει να συγκεντρώνονται όλα αυτά τα στοιχεία και μπορεί τουλάχιστον να εξηγήσει κανείς ε, στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε το αναγνωρίσαμε το πρόβλημα. Πράγματι, η ε, συγκέντρωση δεδομένων θα πρέπει να γίνεται μία και μόνο φορά. Και μία παρατήρηση τώρα προς τους Γάλλους ε, συναδέλφους. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κενά. Εγώ έχω πολύ καλή σχέση προς τον κύριο Σαρκοζή, τον πρώην πρόεδρο. Με τον κύριο Σαρκοζή λοιπόν έχω συζητήσει δυο φορές εκτενώς για το θέμα αυτό. Η Γαλλία δεν έχει τοποθετηθεί επί της ουσίας όσον αφορά ε, στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Όμως στη Μεγάλη Βρετανία το έχουν κάνει κυβέρνηση μπορεί να καταθέσει νόμο μόνο εφόσον καταργεί κάποιον άλλον. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. One in, one out. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ καλό που κάνουν οι Βρετανοί. Οι Σκανδιναβοί και αυτοί προχωράνε. Η Γαλλία όμως, εκεί ε, δεν έχω καταλάβει τη θέση των Γάλλων. Δηλαδή πόσο σοβαρά παίρνει η, κυρίως η νέα γαλλική κυβέρνηση το θέμα της αντιμετώπισης της ε, γραφειοκρατίας. Σας παρακαλώ λοιπόν να το προσέξετε, να ξέρουν οι Γάλλοι ότι ε, πρέπει ε, να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που ακολουθούν οι Άγγλοι, Γερμανοί, οι Σκανδιναβοί, να αντιμετωπίσουν τη γραφειοκρατία ε, και μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά για αυτή την ουσιαστική συζήτηση και σας λέω θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Äh, ευχαριστούμε πολύ κύριε Στόιμπερ. Νομίζω ότι τα χειροκροτήματα είναι απόδειξη του πόσο εκτιμούμε όλοι αυτά που είπατε. Από τότε που είμαι πρόεδρος εδώ στην Επιτροπή αυτή ποτέ δεν είχε γίνει με τόσο ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση. Και πιστεύω ότι χάρη σε εσά και στον τρόπο με τον οποίο ενεργείτε και μας προκαλείτε με αυτά που λέτε, μας κάνετε να σκεφτόμαστε ότι καμιά φορά και εμείς θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και πιο επιθετικοί προς τα έξω και να δείξουμε τι κάνουμε. Νομίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μας αυτό έχουν ως κύριο στόχο. Και δουλεύουν μέχρι εξάντλησης. Καθώς και όλοι οι συνεργάτες της ομάδας μας, όλες τις εβδομάδες είναι εδώ στις Βρυξέλλες, ε, κάνουν ε, τη δουλειά τους ακόμη και τις εβδομάδες που λείπουν οι συνάδελφοι και είναι στις εκλογικές τους περιφέρειες. Πιστεύω όμως ότι μας καταδείξατε με σαφήνεια ότι αυτό που γίνεται και λέγεται εδώ πρέπει και ο τελευταίος πολίτης, ο πιο απομακρυσμένος σε όλες τις χώρες μας να το κατανοεί. Ίσως τώρα με την κρίση του ευρώ θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε τι γλώσσα χρησιμοποιούμε προς τα έξω. Πολύ καλές υποδείξεις μας κάνατε για το θέμα της ε, μεταφοράς της κοινωνικής νομοθεσίας δικής μας που μας αφορά εμάς για το περιβάλλον και μας δώσατε τροφή για περαιτέρω συζητήσεις. Και Καταρχά, ελέγχθη γιατί ένας σοσιαλιστής Γερμανός καλεί έναν πρώην πρόεδρο της Τσεντεού. Το κάνω, το έκανα, διότι στην Επιτροπή και στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών μας παρουσιάσατε, της Τσέσου με συγχωρείτε, ε, παρουσιάσατε κάτι το πολύ ενδιαφέρον και τώρα είδαμε πόσο καλή είναι η εργασία που επιτελείται στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Συνεχίστε με αυτό το ύφο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 θα μας παρουσιάσει το θέμα της, που είναι οι επιλές στο χώρο εργασίας λόγω αμοιάντου και προοπτικές. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν στην ε, έκθεση η οποία κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης, προτάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες. Πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό και ότι λέει δεν είναι χρήσιμο. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στην, στην ε, προηγούμενη θητεία όταν ως κοινοβούλιο ασκήσαμε το δικαίωμα συμμετοχής δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα εμείς για να απαγορεύσουμε κάποια πράγματα. Η νομοθεσία που αφορά την υγεία των πολιτών είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο ε, θέλουμε εμείς να προτείνουμε επιτρέπει τη συμπλήρωση κάποιων στοιχείων ε, της ε, έκθεσης που κάνει η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπής. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα λόγω μεσοφιλιωμάτων και αμυντίου στην Ευρώπη και πολλές επαγγελματικές ασθένειες προκαλούνται από αυτό το λόγο, διότι πάρα πολλοί ε, βρίσκονται σε χώρους οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι πάρα πολύ στο αμύαντο και υπάρχει κίνδυνος. Θα πρέπει να κάνουμε έναν κατάλογο πάρα πολύ λεπτομεριακό, ώστε να μπορέσουμε να επισημάνουμε όλες αυτές τις δυνητικές ε, επιπτώσεις μεσοθυλιώματος ή ε, αμοιάντωσης. Πρόκειται για μια ορολογιακή βόμβα. Όποιοι εργάζονται και ζουν σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ή χρησιμοποιούν τέτοια υλικά έχουν πρόβλημα. Στο 2006 στην εκστρατεία που έγινε ελέγχθη ότι ο αμύαντος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος και όσοι έχουν εργαστεί στην ε, ανακαίνιση έχουν ίσως τα τώρα και δεν θυμούνται που ακριβώ υπήρχε μεγάλη ε, συγκέντρωση. Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και υπάρχει. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα κοινοτικό ταμείο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει πιστούν τέτοιου είδους προβλήματα επαγγελματικών ασθενειών που προκαλούνται από την αμαντίωση. Από ό,τι λέγεται από την Διεθνή Οργάνωση Υγείας υπάρχουν νέα 20 με 30 χιλιάδες περιπτώσεις που, που εμφανίζονται ετησίως και δεν ξέρουμε πού πάμε. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να αυξηθεί το κονδύλι που έχω συμπεριλάβει στη γνωμοδότηση εάν παρουσιαστούν και νέα στοιχεία οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και τα μέλη των οικογενειών των ασθενών θα πρέπει να την χάνουν και κάποιες υποστήριξεις όταν τα πράγματα πηγαίνουν ακόμη και στα δικαστήρια για να επιληθούν τέτοιου πράγματα. Ε, σε μια κρόση που έγινε ζητήσαμε να γίνουν κάποια πράγματα και θέλουμε να ζητήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλους τους υπευθύνους να προβλέψουν κονδύλια για να απαγορευτεί η χρήση του αμοιάντου. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε μέτρα εξυγίανσης στα ήδη υπάρχοντα κτίρια και επίσης ε, ε, τη εξυγίανση των χώρων συμπεριλαμβανομένων και των επισφαλών χώρων υγειομικής ταπείνων αποβλήτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα τελειώνοντας την εταιρεία Eternit και πρέπει να πω ότι άρχισε πήγε υπόθεση στα δικαστήρια το 2009 ο Ελβετός ιδιοκτήτης και διευθυντής κρίθηκαν ένοχοι και ήταν υπεύθυνοι για το περίπου 3.000 θανάτους που σχετίζονται με τον αμύαντο και χρειάστηκε να καταβάλουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων. Τα χρήματα κατεβλήθηκαν στα θύματα, στις οικογένειές τους και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και η δίκη έτερνη εξαιτία της μεγάλης έκταση των θυμάτων θεωρήθηκε η δίκη του αιώνα. Δεδομένου ότι είχαμε να κάνουμε με 3.000 θανάτους από ε, αμοιάντωση και ε, καρκίνο εξαιτίας μεσοφιλιώματο και με πάρα πολλούς ασθενείς. Ευχαριστώ. Das Wort, Eleni το λόγο στην κυρία Θεοχάρη. Έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αμίαντο και γι' αυτό το λόγο είμαι shadow σε αυτό το, το opinion που γράφει η Επιτροπή μας. Ε, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε η εξαιρετική συνάδελφος ότι δεν μπορούμε να την δούμε μόνο ως επαγγελματική νόσο την το ότι προκαλεί ο αμύαντος και την ασβέστωση και το μεσοθυλίωμα και ενδεχομένως το μικροκυταρικό καρκίνωμα. Δεν υπάρχουν ικανοποιητικά επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα που να το καθορίζουν μόνο αυτό το, αυτό το ζήτημα. Πρέπει να το δούμε ως κάτι που αφορά τον γενικότερο πληθυσμό και προς αυτή την κατεύθυνση θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, πανευρωπαϊκή τεκμηριωμένη μελέτη που θα χαρτογραφήσει τις περιοχές της Ευρώπης που υφίστανται αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα και τις ε, συνέπειες του και να ε, ληφθούν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις επιμέρους κοινότητες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να σταματήσει η, εφαρμογή του η χρήση του αμοιάντου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να αναφερθώ ειδικά στην Κύπρο που είναι μια περιοχή η οποία έχει υποστεί πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες. Πρόσφατα υπήρχε μια συζήτηση στην ε, κρατική δανέζικη τηλεόραση, την τηλεόραση της Δανίας, όπου κατηγορήθηκε η εταιρεία FL Smith, η οποία για 80 περίπου χρόνια εκμεταλλευόταν το μεγαλύτερο αμυαντορυχείο σε κάποια φάση της Ευρώπης στην Κύπρο, ότι γνώριζε τις επιπτώσεις πάνω στους εργαζόμενους και στο γενικό πληθυσμό και παρόλα αυτά το άφησε το μεταλλείο να δουλεύει για τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάρθει καμία ε, μα καμία ε, προστασία του γενικού πληθυσμού. Και τώρα, εδώ και 25 χρόνια έχει κλείσει το μεταλλείο, καταμετρούμε πολλούς θανάτους μεσοθυλιώματος σε όλα τα γύρω χωριά. Επιπλέον, η Κύπρος υποφέρει γιατί χρησιμοποιήθηκε ο αμίαντος για τους, για τους σωλήνες της ίδρευσης, για την ε, υδροδότηση ολόκληρου του νησιού. Και παρόλο που υπήρξαν κάποια κοινοτικά κονδύλια και αντικαταστάθηκαν όλοι οι δροσολίνες στις κατεχόμενες περιοχές, στις ελεύθερες περιοχές του νησιού μας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται αμυαντοσολίνες. Δεν υπάρχει καμιά επιστημονική συσχέτιση ακόμα της, ε, του καρκίνου του στομάχου με, την, ε, με τον αμύαντο. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο και πρέπει να ληφθεί και αυτό το φαινόμενο, το, το, η παρατήρηση πάρα πολύ σοβαρά. Διαφορετικά γιατί αντικαταστάθηκαν οι σωλήνες αμοιάντου στις ε, κατεχόμενες περιοχές με κοινοτικά κονδύλια. Επίσης υπάρχει ένας εγκαταλελειμμένος ε, οικισμός των Βρετανικών βάσεων μέσα σε κατοικημένη περιοχή που αποτελείται αποκλειστικά από σπίτια κατασκευασμένα από αμίαντο. Όλα αυτά εκθέτουν τον γενικό πληθυσμό σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Πολλοί προσφυγικοί οικισμοί στις ελεύθερες περιοχές έχουν σπίτια κατασκευασμένα από αμίαντο και επιπλέον έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, ένα ναυάγιο έξω από το λιμάνι της Λεμεσού με χιλιάδες τόνους αμιάντου. Για αυτούς τους λόγους και γνωρίζοντας ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι μόνο η Κύπρος έχει αυτό το, αυτό το ζήτημα, έχει κάνει μια νομοθεσία που απαγορεύει την χρήση του αμοιάντου στα φρένα των αυτοκινήτων σε οικιακά σχέδια ως μονοτικό υλικό, αλλά αυτό δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του μείζωνος προβλήματος της ε, έκθεσης ακόμη σε ενεργείς ίνες του πληθυσμού και της χρήσης των υδροσολύνων και των ε, σπιτιών, θα πρέπει στοχευμένα και στη βάση της γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής που δεν θα δημιουργήσει επιβάρηση του προϋπολογισμού, δεν θα προκαλέσει αντιδράσεις αλλά επιπλέον θα βοηθήσει στην αναστολή της ύφεση στην αντιμετώπιση της ανεργίας να ληφθούν εκείνα τα μέτρα που θα τεκμηριώσουν την, ε, επιστημονική, ε, επιστημονικά την, ε, τις επιπτώσεις του αμοιάντου όχι μόνο ως επαγγελματικής νόσου και θα βοηθήσουν και στην εξάλληψη του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Vielen Ευχαριστούμε πολύ. Η Λίντα Μακέιβαν εκπροσωπεί την ε, ε, σκιώδη συγγήτρια για, το, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Η Γκλένης μου άφησε το ακόλουθο μήνυμα. Θέλει καταρχάς να, βοηθεί, να ευχαριστήσει τη Σαμπίν Βίλς για την πολύ καλή αυτή γνωμοδότησή της, που πραγματικά ελπίζει να βελτιώσει την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος τροπολογίες θα ήθελε να υποβάλει στα εξή σημεία. Καταρχάς την ίδια την ονομασία της έκθεσης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, όπως ακριβώς είπατε κυρία Θεοχάρους, για μια επαγγελματική ασθένεια. Πρόκειται πραγματικά για μια περιβαλλοντική, θα λέγαμε, ασθένεια, που πειράζει πολύ περισσότερους ανθρώπους. Πιστεύει λοιπόν η Γκλένης ότι θα πρέπει να μιλάμε για γενικότερα τις απειλές στην υγεία από τον αμίαντο και όχι μόνο την υγεία στο χώρο της εργασίας. Και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε πολύ, πιστεύω. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να απαγορεύεται η χρήση αμοιάντου και ότι θα πρέπει να προβλεφθεί και μία προθεσμία 2023 συγκεκριμένα, να είναι αυτή η τελική προθεσμία, στην οποία δεν θα δεν θα προβλέπετε, με καμία άλλη εξαίρεση ή προκειμένου να καταργηθεί η χρήση του αμιάντου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. το προβλήμα του αμοιάντου έχει προκαλέσει πάρα πολλούς ε, θανάτους ε, στην Ευρώπη ε, και θα προκαλέσει και άλλους τόσους στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο να μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Λίγες μόνο ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν μεσοτηλίωμα και 40 χρόνια μετά την χρήση του αμοιάντου. Στην Ιταλία υπάρχουν ολόκληρες ολόκληρα κημητήρια ε, τα οποία έχουν ε, νεκρούς λόγω αυτού του προβλήματος. Αν λοιπόν θέλουμε να αποφύγουμε και νέες ε, περιπτώσεις θα πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση αμοιάντου και στα σπίτια και στα εργοστάσια. Πολλές επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι το κόστος όμως είναι απογορευτικό σε μια περίοδο κρίσης γιατί μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά αμοιάντου που θα πρέπει να αντικατασταθούν. Επίσης από την εισηγήτρια έγινε λόγος για αυτή την επιχείρηση στο Τωρίνο και ισχυρίστηκε η εισηγήτρια ότι η επιχείρηση αυτή ήξερε πολύ καλά τον κίνδυνο. Διερωτώμε λοιπόν δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιήσουμε ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς έτσι ώστε όποιος ε, κοινεί ε, προϊόντα που είναι επικίνδυνα ας πούμε στα αυτοκίνητα να είναι να τα αποσύρει. Ε, νομίζω ότι εφόσον γνώριζαν ότι είναι επικίνδυνος ο αμύαντος θα έπρεπε να επιβληθούν οι απαραίτητες κυρώσεις που προβλέπονται για καρκινογενή προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν να περιοριστεί το ανώτατο όριο των ινών που προβλέπεται αυτή τη στιγμή από την νομοθεσία. Γιατί σας είπα, δεν υπάρχει ένα όριο από το οποίο και μετά να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως ε, αυτές οι είναι σε αμοιάντου ε, είναι υπό γίνονται διάφορες εξετάσεις στην Ευρώπη για να μπορεί κανείς να αποφύγει τον κίνδυνο. Στο δικό μας λοιπόν, ε, σε εμά στην Ευρώπη, γίνονται πάρα πολλά για την ε, αντικατάσταση του αμοιάντου και για τα απόβλητα. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλοί χώροι υγιεινής ε, ταφής, πολλές είναι επικίνδυνες. Εγώ ας πούμε ζω σε μια περιοχή 22.000 κατοίκων, όπου έχουμε τέσσερις χώρους υγειονομικής ταφής αμοιάντου. Ο κίνδυνος λοιπόν μόλυνσης από αυτούς τους χώρους υγειονομικής ταφής είναι πάρα πολύ ψηλός. Γιατί εντωμεταξύ ε, έχουν ε, διεισδύσει, είναι σαμιάντου στον υδροφόρο ορίζοντα και ε, αυτές λόγω της διοχέτευσης του νερού και της χρήσης του γενικότερα και στην γεωργία οι σε αυτές από το υπέδαφος τελικά φτάνουν γενικότερα στην ατμόσφαιρα μέσω της άρδευσης και με πολλούς άλλους τρόπους. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει νομοθετικά να ρυθμίζονται ειδικέ χωματερές, ειδικοί χώροι γενομικής ταφής αποβλήτων αμοιάντου. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, το πρόβλημα του ενταφιασμού, της απομάκρυνσης των αποβλήτων, ενέχει κι άλλον ένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ο εξής ο αμίαντος ε, που είναι μια λέξη as best ε, προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και κατ' ουσίαν σημαίνει δεν μπορεί να ε, διαλυθεί. Δεν είναι λοιπόν σωστό τον αμίαντο να τον ενταφιάζουμε στο υπέδαφος. Όχι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία εκείνη που υπάρχει για την απομάκρυνση των αποβλήτων του αμιάντου. Θα πρέπει λοιπόν να αντιρωτηθούμε το εξής. Είναι σωστό να αφήνουμε αυτές τις ε, κατ' ουσίαν βόμβες. Γιατί δεν αποκλείουμε το γεγονός ότι μετά από 200 ή 300 χρόνια ε, θα έρθει κάποιος ο οποίος πάνω από αυτές τις ε, χωματερές θα κατασκευάσει οτιδήποτε, ένα κτίριο ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα και ως εκ τούτου θα πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτούς τους ε, ανοιχτούς χώρους ε, ταφής. Γιατί κατά κάποιον τρόπο είναι μια διαθήκη που αφορά τις επόμενες γενιές. Σε αυτές κληροδοτούμε το πρόβλημα, το οποίο όπως είδαμε πάρα πολύ καλά είναι πολύ οξύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ καλό θέμα στο οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο η Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα για να ενημερώσει, να αλλάξει να προστατεύσει και να απαγορατεύσει. Δεδομένου ότι για χρόνια υπάρχει τέτοιου είδους συνενοχή μεταξύ άλλων, μόνο το 97 απαγορεύτηκε και περιμένουμε τα επόμενα χρόνια στο 2030 100.000 θανάτους. Ε, δεν είναι 25.000 όπως λέει η συγγήτρια. Μέχρι το 2030 θα έχουμε ίσως και 500.000. Και όπως είπε ο κ. Μακεβάλ, θα πρέπει σε σχέση και με άλλους εργαζόμενους που είναι σε κοντινές περιοχές την προστασία, όχι μόνο στους εργαζόμενους. Εάν λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Πολωνία, η Γερμανία χρησιμοποιούν ακόμη ε, τον αμιαντούχο χρυσότυλο, θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι μνήμη θα κρατήσουμε από ό,τι γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται με τις ανακαινήσεις. Εάν δείτε σε πόσα κτίρια, σε σπίτια υπάρχει αμύαντος και ο εργαζόμενος και οι γείτονε θα μολυνθούν. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να γίνει σωστή χαρτογράφηση σε όλες τις χώρες ώστε να εντοπίσουμε πού μπορεί να υπάρχει αμύαντος. Υπάρχει το πρόβλημα των αποβλήτων και υπάρχει και το πρόβλημα των πλοίων. Όπως ξέρετε θα υπάρξει κανονισμός ε, τον οποίο θα μελετήσουμε και τα ευρωπαϊκά πλοία, αυτά τα, τα πλοία τα οποία έχουν ευρωπαϊκή σημαίνα ελέγχονται, αλλά όποια έχουν τρίτων χωρών δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Θα πρέπει λοιπόν επίσης και αυτό το πρόβλημα να το εξετάσουμε. Τώρα, πρόληψη για τους εργαζόμενους, δικαίωμα ενημέρωσης και ενημέρωση των επαγγελματιών, διότι υπάρχει και το εξή ερώτημα. Τι κάνουμε με το Ethernet που υπάρχει σε όλες τις στέγες. Υποχρεώνουμε όλους τους ιδιώτες να τις αφαιρέσουν, γιατί ακόμη τον έχουν τον αμύαντο στην ε, ε, στέγη τους. Τώρα, για τα θύματα, θα ήθελα να υπάρχει εναρμόνιση, διότι κάποιες χώρες λαμβάνουν υπόψη τι ασθένειε και τι θεωρούν επαγγελματικέ ασθένειε. Υπάρχουν όμω άλλε, όπου τα πράγματα είναι ακόμη πολύ πιο δύσκολα. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με ενίσχυση στα θύματα ώστε να δίδονται οι σωστέ αποζημιώσει. πρέπει να σκεφτούμε τα άτομα τα οποία υπέστησαν ότι παίζαν και χωρί να το ξέρουν. Ευχαριστώ, κύριος Σαμπανό. Pane Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή και για την όλη συζήτηση που μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχουμε. Σίγουρα ο αμίαντος αποτελεί μια τεράστια απειλή για την υγεία Φαίνεται ότι δυστυχώς όμως δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ευρωβουλευτές καθότι είμαστε νομίζω μόνο 7 οι οποίοι συμμετέχουμε. Πολλοί δεν φορούν καν τα ακουστικά τους, φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Παρ' όλα αυτά θα πω αυτά τα οποία έχω να πω. Συμφωνώ και εγώ ότι ο αμίαντος δεν αποτελεί απειλή μόνο της υγείας στο χώρο της εργασίας. Είναι μια πολύ ευρύτερη τραγική απειλή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε ένα κείμενο πολύ πιο δυνατό, ένα κείμενο με πυγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταδεικνύεται στο κείμενο αυτό ο πραγματικός κίνδυνος που απορρέει από τη χρήση του Και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσω του κειμένου αυτού να καταφέρουμε να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα επιτόπου. Το ζήτημα του αμίαντου θα απασχολήσει προφανώς και την Επιτροπή Απασχόλησης ως καθήλυνα αρμόδια και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη τα οποία πραγματικά επιθυμούν να έχουν μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για το πώς θα, πώς θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τη χρήση αμοιάντου και πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ευέλτιστες πρακτικές. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι ε, οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμοιάντου μπορούν να καταπολεμηθούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κράτους μέλους, μέσω εθνικής νομοθεσίας. Καθότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια νομική βάση για να εγκριθεί κοινοτική νομοθεσία επί του αμοιάντου. Η Επιτροπή Απασχόλησης στην δική της την έκθεση έχει παραθέσει κάποιες πολύ φιλόδοξες προτάσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά την άποψή μου την αρχή της επικουρικότητας. Σίγουρα θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο του αμοιάντου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσετε να πάρω το λόγο. Ο κύριος Ρώση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω το ζήτημα του αμοιάντου είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να δοθεί εύκολα μία λύση. Ο αμύαντος πάντω προέρχεται από φυσικά υλικά. Εγώ προέρχομαι από το Πιεμόντε και υπάρχει ένα ορυχείο στην περιοχή του Τωρίνου από το οποίο πραγματικά παίρνουμε αμίαντο. Όλε οι γύρω περιοχέ είναι γεμάτε με φυσικό αμίαντο και η περιοχή αυτή η οποία βρίσκεται κοντά στο Ρήνο καθώς επίσης και έργα που γίνεται κοντά στη Λιόν έχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία περιέχουν αμίαντο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέσουμε λοιπόν ανώτατα όρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε τον αέρα, έχουμε τα νερά, που μεταφέρουν ίνες αμιάντου στις γύρω περιοχές. Ακόμα και οι ίδιοι οι γεωργοί όταν καλλιεργούν τη γη τους πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με πολύ υψηλά επίπεδα μιάντου και αυτοί μέσω της καλλιέργειας της γης συμβάλλουν στο να επεκταθούν ακόμα περισσότερο οι ίνες αυτές. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα λοιπόν αυτό πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το ζήτημα της ταφής. Δεν θα πρέπει να μας φοβίζει η ταφή, η γενομική ταφή. Πολύ καλύτερα ο αμύαντος τελικά είναι θαμένος παρά να είναι στην επιφάνεια της γης. Όταν είναι στην επιφάνεια της γης κυκλοφορεί πολύ ελεύθερα. Αν μη τι άλλο όταν είναι θαμένος εκεί πέρα είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Ναι, σίγουρα μπορεί να περάσει ακόμα και στους υδατοφόρους ορίζοντες, αλλά ξέρετε ότι ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αμιάντου ήδη πάνω στις πλαγιές των βουνών του Πιεμόντε. Μόνο και μόνο μέσω της βροχής ο αμίαντος ουσιαστικά μεταφέρεται. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τελικά ο αμίαντο, ο οποίο βρίσκεται μέσα στου σωλήνε των υδραγωγείων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που πίνουν νερό από το σύστημα το οποίο έχει τους σωλήνες αυτούς ουσιαστικά λαμβάνουν άμεσα τον αμίαντο. Ξέρετε ότι το να πίνει κανείς ή ε, να το χρησιμοποιεί το νερό το οποίο περιέχει αμίαντο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα φαινόμενα καρκίνου. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για να μην δαπανίσουν τελικά χρήματα τελικά χρησιμοποιούν, παίρνουν κομμάτια μία του τα οποία τα πουλάνε τελικά μέσα στα ποτάμια. Πάλι στη δικιά μου την περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά πάρα πολύ αμύαντος ουσιαστικά, ο οποίος έχει πεταχτεί ακριβώς μέσα στα, ποτάμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες, να μην προχωρούν σε τέτοιες δραστηριότητες, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να περιορίσουν τη χρήση του αμοιάντου, να επιβάλλουμε ουσιαστικά στα κράτη-μέλη να επέμβουν προκειμένου να αφαιρέσουν τον αμίαντο όταν βρίσκεται σε σημεία που τον καθιστούν ακόμα πιο απικίνδυνο. Σας λέω ότι στο Πιεμόντε έχουμε πραγματικά εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα όπου, στα οποία βρίσκουμε τελικά αμίαντο ο οποίος έχει διατεθεί με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Δεν είναι σωστά διατεθειμένος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα μετά από τι ε, διαπιστώσει που έγιναν και τι παρατηρήσει από του διάφορου βουλευτέ. Συμμερίζομαι αυτό που είπατε. Πρέπει να σα πω ε, ότι έχουμε ένα, μια οδηγία που όταν εφαρμόζεται σωστά επιτρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα. Και επίση όταν εφαρμόζεται σωστά η οδηγία στις εθνικές νομοθεσίες, το ίδιο συμβαίνει. Το πρόβλημα του αμοιάντου στους χώρους εργασίας το χειριζόμαστε στο πιο γενικότερο πλαίσιο των επαγγελματικών ασθενειών. Δημοσιεύθηκε πρόσφατα μία έκθεση που υπάρχει στο ίντερνετ και του χρόνου θα έχουμε μία διάσκεψη για τις επαγγελματικές ασθένειες και εκεί θα συζητηθεί επίσης το πράγμα. Αλλά όντως Θα συνεχίσουμε την εργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της έκθεσης αυτής για να δούμε εάν θα πρέπει να συνεχιστούν οι δράσεις μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βίλς, πάρα πολύ σύντομα για να ολοκληρώσουμε. Ναι, Νομίζω ότι ξεπεράσαμε το χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις τοποθετήσεις τους όλους τους συναδέλφους. Χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ όλων η γνωμοδότησή μου θα είναι καλή. Εγώ θα ήθελα να απαγορευτεί η χρήση του αμοιάντου. Αυτό είναι το διατάφτα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, όλους όσους συμμετείχαν στην συζήτηση πρέπει να πω ότι και εγώ πήγα στην Κύπρο και τόπου επισκέφθηκα τις εγκαταστάσεις αυτής και όντως θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, καταστρέφοντας όλες αυτές τις ε, ύποπτες εγκαταστάσεις να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ε, καλή όρεξη. Θα τα ξαναπούμε στις 3 για να συνεχίσουμε και να συναντήσουμε τον κύριο Σπρέγκερ.